Συνάδελφοι, έχουμε ένα πολύ γεμάτο απόγευμα. Θα ξεκινήσουμε με τον Επίτροπο Κάλλος που θα παρουσιάσει την ενδιάμεση αναθεώρηση και μετά έχουμε τους τέσσερις υπολείπους συντονιστές για τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Θα πρέπει να είμαι αρκετά αυστηρός ως προς το χρόνο. Χωρίς λοιπόν πολλά πολλά, να ξεκινήσουμε με τον Επίτροπο Κάλλας. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί βουλευτές, ε, είναι μεγάλη μου ικανοποίηση να παρουσιάσω την ενδιάμεση αναθεώρηση και θα μιλήσω για τα προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από τα διευρωπαϊκά δίχτυα. Οι συντονιστές έχουν ε, συμβάλει ε, στην διάμεση αυτή αναθεώρηση και θα βοηθήσουν να εφαρμοστούν τα αποτελέσματα. Η ενδιάμεση αναθεώρηση θα σας δώσει μια λεπτομερή εικόνα του πού βρισκόμαστε, ε, ιδιαίτερα ως προς ε, τα 30 προγράμματα προτεραιότητας. Ε, καταρχήν θα επικεντρωθώ σύντομα στα διευρωπαϊκά δίκτυα όσα έχουν σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη καταλάβει από κάποιους από τους συντονιστές που βρίσκονται σε κάπως διφορούμενη θέση. Από τη μία μεριά τα κράτη-μέλη καταβάλουν προσπάθειες ε, παρά τις οικονομικές δυσκολίες ε, που αντιμετωπίζουν. Κάποια από τα προγράμματα έχουν καθυστερήσει λόγω έλλειψης πόρων, η εφαρμογή έχει καθυστερήσει, νέα προγράμματα αντιμετωπίζουν προβλήματα στο ξεκίνημά τους καθότι απαιτούν σημαντικές επενδύσεις. Επίσης βλέπω ότι αντιμετωπίζουμε επίσης ε, μια κατάσταση που μοιάζει με patchwork. Είναι πολύ διαφορετικές οι καταστάσεις ε, στα διάφορα κράτη-μέλη και στις διάφορες περιοχές. Είναι λοιπόν πολύ δύσκολο να διατηρήσουμε την ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεγάλο πρόγραμμα είναι η ε, το τούνελ Μπρένερ. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε κατασκευή, όπως και για την γραμμή ψηλή ταχύτητα ε, ε, ε, Μαδρίτη Λισαβόνα. Επίση, χώρε όπω η Ιταλία, οι κάτω χώρε, η Αυστρία και η Δανία έχουμε προγράμματα τα οποία αντιμετωπίζουμε προβλήματα και στη Γερμανία αντιμετωπίζουμε προβλήματα για να έχουμε τα απόλυτα διαλειτουργικά δίκτυα που θέλουμε για να έχουμε μια ε, λειτουργική εσωτερική αγορά στη μεταφορά. Ωστόσο, ε, είμαι αισιόδοξο όσον αφορά την συνεχιζόμενη χρηματοδότηση και ε, καταβολή προσπαθειών. Το 2010 είδαμε ολοκλήρωση κάποιων τμήματων ε, στα οποία είχαμε επενδύσει χρήματα από τα διευρωπαϊκά δίκτυα όπως είναι η σύνδεση υψηλής ταχύτητας Ελιέγης και Άχεν, την γραμμή Στρασβούργου ε, και έχουμε το ε, Περπινιόν ε, Φιγκέρας μεταξύ Ισπανίας και Γαλλίας. Είναι προτεραιότητά μας η διαλειτουργικότητα και στην στο πολιετές ε, πρόγραμμα ε, συλλέξαμε προτάσεις ε, που θα εφαρμοστούν από το 2007 μέχρι το 2013. Τα 92 αυτά προγράμματα αντιπροσωπεύουν τα 2 τρίτα του συνολικού προϋπολογισμού των διευρωπαϊκών δικτύων 5 δισεκατομμύρια κάτι από από 8 δισεκατομμύρια συνολικά μιλάμε για 32 ε, δισεκατομμύρια, 647 εκατομμύρια συνολικά που θα στοιχήσει η χρηματοδότηση των έργων αυτών. Τα προγράμματα αυτά έχουν αναλυθεί λεπτομερώς ε, από εσωτερικούς και εξωτερικούς εμπειρογνώμονες και η ανάλυση αυτή έχει οδηγήσει στην έκθεση που έχετε στα χέρια σας αυτή τη στιγμή. Η έκθεση αυτή δείχνει ότι ο προϋπολογισμός των διευρωπαϊκών δικτύων ε, αποτελεί αντικείμενο πολύ αυστηρής ε, διαχείρισης. Ε, συνεχίζεται η πρόοδος. Είχαμε την επιλογή ανάμεσα σε κάποια προγράμματα τα οποία δεν θα είχαν ολοκληρωθεί μέχρι το 2013. Θα έπρεπε αυτά τα προγράμματα να συνεχιστούν και στι επόμενες δημοσιονομικές ε, προοπτικές ε, Το 2014, 2015, 2016, 2017 ή ακόμα και πιο μετά. Προφανώς αυτός δεν είναι καλός τρόπος διαχείριση του προϋπολογισμού των διευρωπαϊκών δικτύων. Γι' αυτό προτείνω να βρούμε μια ισορροπία να επιτρέψουμε σε προγράμματα να συνεχιστούν για δύο χρόνια παραπάνω, να μην ε, κόψουμε οποιαδήποτε χρηματοδο... να κόψουμε οποιαδήποτε χρηματοδότηση μετά το 2015 και η παράταση αυτή θα δοθεί μόνο υπό αυστηρούς όρους. Ε, οι ε, όροι αυτοί είναι πολιτικής, ε, οικονομικής και τεχνικής φύσης. Η απόφαση αυτή θα επιτρέψει σε άλλα 29 έργα να ολοκληρωθούν, αφήνοντα μόνο το 6% του προπολογισμού που να μην έχει απορροφηθεί επιπλέον. Ε, ο προπολογισμό. Ε, που θα ε, ε, περικοπεί τους επόμενους μήνες θα επανιστρέψει στα διευρωπαϊκά δίκτυα. Πάνω από 300 δισεκατομμύρια ευρώ θα εκατομμύρια ευρώ συγγνώμη, θα δοθούν και θα προγραμματίσουμε τη ρήτρα διακοπής του, της χρηματοδότησης το 2013. Θα υπάρχει και το συνηθισμένο Ντρουάντε Ρεγκάρ. Και όπω ξέρετε, εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ η διαφάνεια και η υποχρέωση λογοδοσία. Η έκθεση αυτή σα δίνει όλε τι σχετικέ λεπτομέρειε. Η αναθεώρηση δεν ήταν εύκολη Ο ε, ε φτωχό προπολογισμό των διευρωπαϊκών δικτύων θα χρησιμοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα μπλοκάρουμε καμία χρηματοδότηση για προ... θα ε, μπλοκάρουμε ε, τη χρηματοδότηση για προγράμματα τα οποία δεν αποδίδουν. Όπω έχω πει, ε, στην περίπτωση χορήγηση παράταση, οι όροι θα διασφαλίζουν την ολοκλήρωση των έργων. Όλε αυτέ οι προποθέσει θα επιτρέψουν περικοπέ στον προπολογισμό και ανακατανομή των χρημάτων. Να σα θυμίσω ότι από τον ε, από τον ε, συνολικό προπολογισμό 8 δισεκατομμυρίων, ε, μόνο 32 ε, εκατομμύρια, λιγότερο από μισό τα 100 δεν έχει δαπανηθεί. Ήδη έχουμε ξεπεράσει το μέσο του διαστήματο αυτού, αντιμετωπίζουμε οικονομικέ δυσκολίε και θα ήθελα λοιπόν να αναφερθώ στι μελλοντικέ δημοσιονομικέ προοπτικέ. Κύριοι βουλευτέ, θα ήθελα να κλείσω με μια ενημέρωση σχετικά με την πολιτική των διευρωπαϊκών δικτύων. Όπω ξέρετε, το δεύτερο έγγραφο διαβουλεύσεων ε, δημοσιεύτηκε φέτος τον Μάιο και παρουσιάστηκε στη διάσκεψη της Ε, Σχεδόν 250 ε, συνεισφορέ λάβαμε από τα κράτη-μέλη, ε, από σημαντικούς περιφερειακούς φορείς, άλλους ενδιαφερομένους και φορείς που αντιπροσωπεύουν περιφερειακές και τοπικές πρωτοβουλίες και προγράμματα. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω τα προγράμματα αυτής της διαβούλευσης. Το ενδιάμεσο αυτό βήμα θα γίνει φέτος ως απαραίτητο βήμα πριν την ε, αναθεώρηση του νέου οδηγού που προβλέπεται να δημοσιευτεί ε, την άνοιξη του 2011. Βλέπω από την αναθεώρηση αυτή ε, να αναδύεται ένα δίκτυο πυρηνικό, κεντρικό και έτσι θα ξεπεράσουμε τα προβλήματα ε, τα διασυνοριακά και διαλειτουργικότητα που ε, αντιμετωπίζουμε. Φαίνεται ότι τα αντιμετωπίζουμε αυτά βήμα προ βήμα και το ε, πυρηνικό δίκτυο θα βασίζεται στη δουλειά των συντονιστών και θα φροντίσουμε οι διάδρομοι να βασίζονται σε μια συνεπή ανάλυση συνεχίσω ε, την δέσμευσή μου για να διατηρήσω τη στενή συνεργασία και προσλέπω ε, στην επόμενη συνάντησή μας ε, για να σας παρουσιάσω τα βήματα αυτά πριν το τέλος του χρόνου. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Τώρα έχουμε του συντονιστές και θα πρέπει να δούμε λιγάκι το θέμα του χρόνου ομιλία. Πώς θα το ρυθμίσουμε. Uh, Οι συντονιστέ, λοιπόν. Τρία λεπτά. Ο κύριος Γκρό, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Καταρχήν σας ευχαριστώ πολύ για τη δουλειά που έχετε κάνει. Το έγγραφο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και η δηλώσεις σας με κάποιες διευκρινήσεις. Πιστεύω ότι θα μπορέσουν ε, να χαρακτηριστούν ε, προσανατολισμένες προς το μέλλον. Ε, το σύστημα αυτό το ξέρουμε εδώ και χρόνια. Ε, καταρχήν είναι θέματα προτεραιότητας, δεύτερον έχουν γίνει πολύ λίγα βήματα πρόοδου και τρίτον δεν υπάρχουν χρήματα. με τα κριτήρια αυτά δεν μπορούμε να διατηρήσουμε ε, τις ε, ίδιες προτεραιότητες, δεν μπορούμε να προσθέσουμε νέες προτεραιότητες και προς τα έξω δίνουμε την εντύπωση ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν είμαστε σε θέση να ολοκληρώσουμε τα ε, προγράμματα αυτά. Πιστεύω ότι είναι πολύ πιο ρεαλιστικό ο τρόπο ο δικό σα να προσεγγίσετε το θέμα. Χρειαζόμαστε λιγότερε προτεραιότητε, χρειαζόμαστε συγκεντρωμένο χρήμα Μπορούμε να δώσουμε παράταση. Χαίρομαι όμως πάρα πολύ που είπατε επίσης ότι η παράταση αυτή των δύο ετών θα συνδέεται με κάποιες προϋποθέσεις. Ε, διότι στα, ε, κατά τη γνώμη μου ε, η πρώτη προϋπόθεση θα πρέπει να είναι ότι το πρόγραμμα έχει ξεκινήσει. Δεν μπορούμε να δώσουμε παράταση δύο ετών για προγράμματα που δεν έχουν καν ξεκινήσει. Έτσι λοιπόν μπορούμε να αποφύγουμε να ε, ε, δεσμεύουμε χρήματα ε, που δεν έχουν απορροφηθεί κάπου όπου δεν θα χρησιμοποιηθούν ούτως ή άλλως. Στο εγγύ μέλλον θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε διασυνοριακά, θα πρέπει να περιοριστούμε σε διασυνοριακά έργα θα πρέπει να, εξετάσουμε, να περιοριστούμε στα bottlenecks που γνωρίζουμε από καιρό τα σημεία συμφόρηση και θα πρέπει να έχουμε συνεπή πολιτική και σε άλλους τομείς ε, πρέπει να συντονιστούμε με την περιφερειακή πολιτική και με την περιβαλλοντική πολιτική. Πιστεύω ότι είναι καιρός στο Κοινοβούλιο μεταξύ των Επιτροπών αλλά και εντός της Κομισιόν να έχουμε πολύ πιο συνεπή προσέγγιση στα προγράμματα αυτά. Αυτό θα ε, ωφελήσει όχι μόνο τη χρηματοδότηση, διότι ιδιαίτερα ε, στο Ταμείο Συνοχής ε, έχουμε πόρους που χρησιμοποιούνται για τα θέματα αυτά, αλλά και για διάφορες περιφέρειες αυτό θα αποτελέσει κάτι θετικό. Εμείς στο ΕΛΚ θα εξετάσουμε προσεκτικά το έγγραφο αυτό και μπορείτε να, βασίζετε, να βασίζεστε σε επικοδομητική συμβολή από το μέρος μας. Προς το παρόν σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας. Ευχαριστώ κύριε Γκρό. Ε, ε, τηρήσατε το χρόνο. Κύριος Αλκαντράου, τρία λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Η αξιολόγηση αυτή που κάνετε μας δείχνει πόσο απαραίτητη είναι μία προσεκτική εξέταση του θέματος. Έχουμε καταλήξει σε ορισμένα συμπεράσματα. Η υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Είναι απίστευτο το 35% των εγγράφων καταφέρνουν να ακολουθήσουν το χρονοδιάγραμμα όπως έχει οριστεί. Αυτό σημαίνει ότι η πλειοψηφία των έργων παρουσιάζει μια καθυστέρηση. προτείνεται μία παράταση δύο ετών για ορισμένα έργα. Ορίζεται όμως μία προθεσμία και συγκεντρώνεται τα μέσα που είναι στη διάθεσή μας. Αυτό είναι απαραίτητο για να μην πάνε χαμένα όλα αυτά τα κονδύλια. Θα επιθυμούσα να γνωρίζω, εάν έχετε ήδη κατά νου ορισμένες προτεραιότητες, προτεραιότητες που θα πετούσαν επιπλέον κονδύλια. Μήπως μπορείτε να μας επιβεβαιώσετε ότι τα έργα αυτά θα συμπεριληφθούν μεταξύ των ε, βασικών έργων. Στον επόμενο προγραμματισμό θα υπάρχουν τα απαραίτητα κονδύλια. Μιλάμε για τον πολιετή προγραμματισμό. Δίκως άλλο, τους επόμενους μήνες θα μπορέσει να γίνει μια συζήτηση για το μέλλον. Θα πρέπει να καθορίσουμε τις προτεραιότητές μας και να κάνουμε επίδειξη μεγαλύτερης δημιουργικότητας για να γίνει μια καλύτερη τοποθέτηση. Θα πρέπει να αξιολογήσουμε τα διαρθρωτικά κονδύλια του Ταμείου Συνοχής, τα οποία θα πρέπει να επαναπροσανατολιστούν και μετά θα πρέπει να βρούμε νέα κονδύλια χρηματοδότηση. Αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση. Τρίτο σημείο, το θέμα του συντονισμού. Πώς είναι δυνατόν να αγγιθούμε μια προστιθέμενη ευρωπαϊκή αξία, έτσι ώστε η Ευρώπη μέσω των συντονιστών να μπορέσει να έχει κάποια βαρύτητα στην ε, αντιμετώπιση και στην εφαρμογή των προγραμμάτων. Εμείς οι σοσιαλδημοκράτες θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να σας βοηθήσουμε να επεξεργαστείτε ένα ολοκληρωμένο δίκτυο. Ε, ευχαριστώ κύριος Μάιστερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ για την παρουσίασή σας και για το έγγραφο που μας ε, δώσατε. Νομίζω ότι όλες ε, οι παρεμβάσεις ε, θα έχουν το ίδιο θέμα, διότι τα, τα προβλήματα είναι γνωστά. Στόχος μας είναι να έχουμε μια εσωτερική αγορά στις μεταφορές. Υπάρχουν όμως και εμπόδια. Και η η Γερμανία όμως είναι χώρα όπου υπάρχουν ε, προβλήματα. Θα πρέπει να δούμε εμείς πώς ε, ως Ευρωπαίοι, ε, ως Ευρωβουλευτές μπορούμε να προωθήσουμε την απελευθέρωση. Μιλήσατε και για τη Σαραγώσα στο μέλλον πώς μπορούμε να βρούμε περισσότερη χρηματοδότηση, πώς μπορούμε να κάνουμε επιλογή των έργων και έτσι φτάνω στην ερώτησή μου που συνδέεται με αυτό που είπατε. Ε, είπατε και πολύ σωστά ότι ε, για την ε, περαιτέρω χρηματοδότηση θα τεθούν πολιτικοί, οικονομικοί και περιβαλλοντικοί όροι. Πολιτικό όρο εννοείται, όταν λέτε πολιτικό όρο εννοείται ότι μπορεί κανείς ε, να αρνηθεί τη χρηματοδότηση σε μια χώρα αν δεν μπορεί να προχωρήσει κάποια ε, έργα. Για παράδειγμα, Ακούσαμε για παράδειγμα ε, σήμερα το πρωί ότι στη χώρα σας πάνε πολύ καλά τα πράγματα αλλά στην ε, Λιθουανία και στην ε, Λετωνία δεν πάνε πολύ καλά τα πράγματα. Μπορεί λοιπόν να λείπουν σε κάποιες χώρες σιδηροδρομικές γραμμές. Μπορείτε λοιπόν εσείς να πείτε ότι πολιτικός όρος είναι να υπάρχει παντού λειτουργικό σιδηροδρομικό δίκτυο και ακόμα και όταν τα κράτη-μέλη δεν είναι σε θέση να χρηματοδοτήσουν τότε θα βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη ή θα πείτε ότι μόνο όπου μπορούν να συγχρηματοδοτήσουν τα κράτη-μέλη θα συνεισφέρουμε κι εμείς που είναι η παρούσα πολιτική μας. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κράμερ, τρία λεπτά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και εγώ για την έκθεση αυτή. Πιστεύω ότι ε, τα όσα ακούσαμε σήμερα ε, θα αποτελέσουν, ε, η σημερινή συνάντηση θα αποτελέσει προηγούμενο. Εξετάζουμε τι δεν έχει πάει πολύ καλά, θέτουμε όρους και ρωτάμε, εξετάζουμε γιατί δεν έχουν προχωρήσει τα πράγματα. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι καλό το ότι σήμερα μπορούμε να συζητήσουμε τα θέματα αυτά. Ο κύριος Γκρός είπε ότι τα διασυνοριακά έργα και τα σημεία συμφόρηση, τα bottlenecks, θα αποτελέσουν ε, ε, προτεραιότητε. Εάν όμω θέσουμε νέε προτεραιότητε, ε, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι κάπου αλλού θα πρέπει να κόψουμε από κάπου αλλού. Και το κέντρο βάρου είναι τα εθνικά προγράμματα. Εάν ε, στη Γερμανία ε, ε, υλοποιηθεί το πρόγραμμα του 21 και στο δάσο του Ριγγίας το σχετικό πρόγραμμα, τότε θα έχει ήδη εξαφανιστεί το 80% της χρηματοδότησης για τα επόμενα 10 χρόνια. Γι' αυτό θα πρέπει να επικεντρωθούμε, θα πρέπει να δούμε πού δαπανείται το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων από τα τέσσερα μεγαλύτερα προγράμματα ε, της ε, Ευρώπης, από τα τέσσερα μεγάλα προγράμματα, τα τρία είναι με ιταλική ε, συμμετοχή. Δεν έχουν όμως σχέδιο χρηματοδότησης. Θα κάνουμε γι' αυτό. Θα γλιτώσουμε πολλά χρήματα εάν λάβουμε σοβαρά υπόψη τους όρους που αναφέρετε εσείς. να πούμε ότι τέρμα το έργο της Μεσίνα, τέρμα ε, το, ε, το, η σύνδεση Λιών ε, Τουρίν, διότι χρειαζόμαστε αλλού τα χρήματα. Νομίζω ότι αυτό είναι απόλυτα ειλικρινές και θα πρέπει να το καταλάβουν οι άλλοι. Επίσης ε, συμφωνούμε με τα όσα είπατε που συμφωνήθηκαν στην Σαραγώσα ε, και όλα αυτά περιλαμβάνονται στην έκθεση της Εύα Λίχτενπέργκε. Θέλουμε νέες προτεραιότητες, θέλουμε να καταπολεμήσουμε τα σημεία συμφόρησης. Αυτά θα πρέπει πρώτα να λυθούν και κατόπιν να ε, προχωρήσουμε σε νέες διαδρομές. Και τελευταίο σημείο που θα ήθελα να αναφέρω. Υπάρχει αντίσταση από τον πληθυσμό. Λιόν Τουρίν για παράδειγμα. Έχετε λάβει σχετική έκθεση και εμείς την έχουμε λάβει. Θέλετε να επιμείνετε παρά τις αντιθέσεις. Η Στουτγκάρδη 21 ε, είναι πρόγραμμα ε, που αφορά όχι μόνο την ε, περιφέρεια της Στουτγκάρδη, αφορά και τη Γερμανία και την Ευρώπη. Πώς θα αντιμετωπίσετε το θέμα αυτό και το τρίτο εμπόδιο είναι η έλλειψη συμμετοχής των κρατών μελών. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε εμείς εάν ένα κράτος μέλος δεν θέλει να προγραμματοποιήσει ένα έργο. Ό,τι και να κάνουμε, κολοτούμπες να κάνουμε, δεν θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα. Γι' αυτό θα πρέπει να δούμε πώ μπορούμε να ε, αντιμετωπίσουμε τα τρία αυτά εμπόδια. Τελευταία παρατήρηση, πολύ σύντομα. Κατά την κατανομή των χρημάτων, κατά τη συγχρηματοδότηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, τα μεγάλα ε, προγράμματα παίρνουν άνετα 25% συγχρηματοδότηση. Άλλα έργα όμω, όπω η σιδηροδρομική γραμμή τη Βαλτική, το Rail Baltica, παίρνουν μόνο 10%. Μήπω μπορούμε και εδώ πέρα να αλλάξουμε τι προτεραιότητε. Ευχαριστώ πολύ. Thank Ωραία. Για τα υπόλοιπα μέλη, δύο λεπτά. Κύριε Καντσάνη, έχετε δύο λεπτά στη διάθεσή σας. Αμέσως ξεκινάω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε που καταφέρατε να κάνετε μία θαυμάσια δουλειά ανακεφαλαιώνοντας ε, όλα τα έργα και ελπίζω να έχουμε τη δυνατότητα να μπορέσουμε να τα ξανακοιτάξουμε. Δεν κατάφερα να τα εξετάσω όλα. Παρ' αυτά παρατήρησα το εξή. Το πρόβλημα των καθυστερήσεων, κύριε Επίτροπε, είναι ένα θέμα. Υπάρχουν, ε, υπάρχει γραφειοκρατία, υπάρχουν τοπικέ πολιτικές. Υπάρχει όμως και το κόστος συγχρηματοδότηση που δυστυχώ ε, σήμερα είναι το πραγματικό πρόβλημα. Δεν είναι λοιπόν μόνο μία απλή καθυστέρηση είναι παράδοξο το γεγονό ότι μπροστά σε μια κατάσταση κρίση με την οποία βρισκόμαστε αντιμέτωποι, μπροστά φτάμε σε μία, ε, σε μία περίοδο ανεργίας, εμείς συσσωρεύουμε καθυστερήσεις σε περιοχές από που περνάνε αυτοί οι διάδρομοι. Είμαι πεπισμένος ότι το να υιοθετήσουμε μέτρα ή να αποχρηματοδοτήσουμε δεν είναι ότι συμβαίνει παρέμβαση σε αυτή την περιοχή, σε αυτή τη χώρα. Απλά και μόνο μπλοκάρουμε ένα διάδρομο και πραγματικά με εκπλήσει το γεγονό ότι στην ε, αναθεώρηση συζητάμε το θέμα της εφαρμοσιμότητας, ε, του, ε, της προτεραιότητας 6-7 ε, το, το, το 1 ή το 6. Αυτό σημαίνει ότι κάνουμε κα, βήματα πίσω σε σχέση με 20 χρόνια προγραμματισμού. Ε, δεν είναι σωστό να κάνουμε ένα βήμα μπροστά και μετά να κάνουμε βήμα πίσω. Καθορίζουμε τις προτεραιότητες Ό,τι ήταν να γίνει, έγινε. Προχωρήσαμε σε επίπεδο σχεδιασμού και αν δεν έγινε το Μπρένερο, Αν δεν έγιναν πράγματα σε τοπικό επίπεδο, είναι προβλήματα που θα πρέπει να λυθούν γιατί υπάρχουν και πολλά έργα που τελείωσαν. Δεύτερο θέμα δεν θα πρέπει αυτό να έχει επίπτωση στη χρηματοδότηση γιατί θα μπλοκάρει τις, ε, τους διαδρόμους. Καλή η παράταση μέχρι το 2015. Σε ό,τι αφορά την εφαρμογή θα πρέπει να κάνουμε αυτή τη σημαντική προσπάθεια στην οποία αναφερθήκατε και ο κύριος Μπαρόζο και εσείς. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λεμπράτσκι, δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, όπως είπε μόλις ο κύριος Αλκαντράουι, και εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να σας συγχαρώ για όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα. Και σε σύγκριση με άλλα έργα, πιστεύω ότι τα διευρωπαϊκά δίκτυα τα πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Ένα-δύο σχόλια, κύριε Επίτροπε. Μήπως θα έπρεπε να γίνει μία, ένα συσχετισμό μεταξύ των ε, κονδυλίων του Ταμείου Συνοχής. Θα ήθελα να γνωρίζω κάτι περισσότερο σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται τα κονδύλια στις χώρες μέλη για το TNT. Γιατί θα πρέπει να βρούμε τι καθυστερήσεις έχουν καταγραφεί σε ό,τι αφορά την, ε, ε, το TNT. Ε, δεν θα πρέπει να επικεντρωνόμαστε μόνο στα, έργα στις πιο πλούσιες χώρες της Ευρώπης. Θα πρέπει να συνυπολογίζουμε και τις χώρες εκείνες που πρόσφατα εντάχθηκαν την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί ενδεχομένω εκεί βρίσκονται τα προβλήματα. Να κάνουμε... Η κυρία Σάβησα, ευχαριστώ πολύ. Ήταν πολύ καλή αυτή η γενική παρουσίαση που μας κάνατε. Και επειδή οι συντονιστές ε, στάθηκαν στα πιο γενικά ζητήματα, θα ήθελα εγώ να σταθώ στις λεπτομέρειες. Σαφώ πάντα όλοι θέλουμε να συζητάμε θέματα τα οποία μα ενδιαφέρουν ιδιαίτερα. Εγώ θα ήθελα να μιλήσω για το δικό μου αγαπημένο πρόγραμμα, το σιδηρόδρομο τη Βαλτική. Σήμερα το πρωί ακούσαμε τον κύριο Μπότσκα να λέει ότι είναι πολύ ικανοποιημένο με την πρώτη φάση του σχεδίου, αλλά δεν πάβει να είναι το πρώτο στάδιο αυτό. Επίση μα είπε ότι θεωρεί ότι είναι προφανέ ότι θα υπάρχει ένα καθημερινό τρένο το οποίο θα πηγαίνει από το Τάλιν ε, στην ε, ε, Βαλτική και πίσω. Ε, το θέμα είναι ε, τι θα κάνουμε. Θα χρησιμοποιήσουμε την ε, Ευρωπαϊκή Οδό, θα χρησιμοποιήσουμε άλλη οδό. Το συζητήσατε εσείς αυτό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι η μία μέθοδος είναι πολύ πιο ακριβή από την άλλη. Και εσείς φυσικά καταλαβαίνετε ε, διαφορετικά πώς έρχονται τα πράγματα. θα περάσετε επίσης στην Εστονία από, την, από τον Πέρνο ή από τον Βάλγκα. Θα πρέπει να επιλέξετε και τις πόλεις εκεί. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο Κάλλας ε, για την παρουσίασή του. Επειδή ο πρόεδρος ε, μας ε, περιμένει με το τσεκουράκι, θα τηρήσω το χρονοδιάγραμμα. Καταρχάς να σας συγχαρώ γιατί είστε αισιόδοξο. Μακάρι όμως, μακάρι αυτή η αισιοδοξία να μεταφραστεί σε έργα. Ε, αναφέρεστε στη λύση κάποιων διαμεθοριακών θεμάτων και αναφέρεστε στο Περπινιάν Φιγκέιρας σας συγχαίρω, αλλά δεν ξέρω κατά πόσον ε, αυτά τα προγράμματα ε, μπορούν να προχωρήσουν. Μία παράταση δύο ετών για τα προγράμματα τα οποία ε, φαίνεται ότι έχουν προχωρήσει καλά και θα ολοκληρωθούν είναι καλή λύση και σας συγχαίρω. Επίσης θα πρέπει να δούμε και τι γίνεται με τα προγράμματα τα οποία δεν είναι βιώσιμα. Θα πρέπει να γίνει ανακατανομή των πόρων μας. Είπατε σωστό, συμφωνώ και με αυτό. Θα ήθελα όμως να σας πω και το εξής. Σήμερα ο κύριος Σαβαρή όταν ε, παρουσίαζε το πρόγραμμά του, μας είπε, ομολόγησε ότι υπάρχουν κάποιες χώρες οι οποίες δεν έχουν πόρος ε, για τα διευρωπαϊκά δίκτυα και θα πρέπει να θέσουν ε, διαφορετικές προτεραιότητες για τις εθνικές τους ανάγκες. Είναι απόλυτα δεκτό αυτό Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να μιλήσετε με τις ε, χώρες μέλη και με τις ε, κυβερνήσεις για να δείτε ποιο είναι διατεθειμένος και ποιο έχει και πόρου για να αντιμετωπίσει το θέμα και από πολιτική αλλά και από οικονομική πλευρά με σύμπραξη ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και τι μπορεί να γίνει βάσει αυτών των πόρων. Να σας πω το εξή. Ε, ο διάδρομος της Μεσογείων. Ε, εγώ καταλαβαίνω ότι με τον έλεγχο θα είναι υπέρ, δεν ξέρω κατά πόσον θα είναι βιώσιμο, αλλά εγώ δεν θέλω να είναι κατά οποιοδήποτε προγράμματος. Υπάρχει όμως ε, ένα πρόβλημα και ελέγχοντας τις χώρες μέλη θα πρέπει να δούμε ποιοι μπορούν να χρηματοδοτήσουν και να υποστηρίξουν προγράμματα τα οποία θα έχουν την ίδια βιωσιμότητα. Ευχαριστούμε τον κύριο Γκράντε Πασχουάλ. Ο κύριο Γκράντε Πασχουάλ έχει δίκιο. Είμαι πολύ αυστηρό με το χρονοδιάγραμμα γιατί έχω άλλου 10 στον κατάλογό μου. Γι' αυτό λοιπόν δύο λεπτά ο καθένα. Η κυρία Γιάλα Σέντερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Κάλλας, Εγώ δεν θα ακολουθήσω τη διαδικασία σας, διότι με εκπλήσει το γεγονός ότι ξεκινώντας από έναν ε, προϋπολογισμό του 2007-2013, ο οποίος ε, είναι κατακρεουργημένος και που άλλοι επίτροποι πήραν πολύ περισσότερα από ό,τι ε, με εκπλήσει όλη αυτή η διαδικασία. Σε καμία από τις προηγούμενες διακουλεύσεις, σε καμία από τις άλλες ομάδες χρηματοδοτήσεις δεν είχε προκύψει μια τέτοια πρόταση. Ουσιαστικά έχουμε μια μεταφορά των διαθροτικών κονδυλίων. Μου δίνεται εντύπωση ότι το μήνυμα που δίνουμε προς τα έξω είναι ότι παρετούμεθα πριν ακόμα ξεκινήσει η συζήτηση. Ε, και δεν θα έχουμε πόρους για τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Τι κάνουμε, θα έχουμε μόνοι μας την ίδια μας υπόθεση. Είναι πολύ εντυπωσιακό το γεγονός ότι αλλάζουμε την τοποθέτησή μας στα μισά του δρόμου. Ούτε το Γαλιλαίο προχώρησε, ούτε τίποτα άλλο όταν κάναμε τέτοιου τύπου αλλαγές. Επομένως δεν καταλαβαίνω τι γίνεται όταν αρχίζουμε να κάνουμε διαφορετικές ε, προσανατολισμούς χωρίς να έχουμε εξοισορροπήσει τα πράγματα, να δούμε τι γίνεται με τις περιφέρειες, με τις ε, θέσεις εργασίας, με τις ε, με οτιδήποτε. Το να πούμε ότι θα παλέψω για να πετύχω αυτό αρκεί να μπορέσω να πετύχω το σωστό αποτέλεσμα, ε, ναι, μεν δεκτό, αλλά το να τα περικόψουμε ξαφνικά είναι σαν να λέμε ότι δεν λειτουργούν τα διευρωπαϊκά ε, δίκτυα, καθυστερούν, δεν είναι σοβαρά και μάλιστα υπάρχουν πολλά προβλήματα και όπως έλεγε και ο συνάδελφος, ε, ουσιαστικά σταματάμε διαδικασίες όπως το Μπρένερο, το, ε, Ταλής ε, τα νέα προγράμματα, τε, Βόρεια Παλμέγια Βάλκα, καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν μια σειρά από προγράμματα. Υπάρχει και το πρόγραμμα PP16 που δεν προχωράει στην ε, περιοχή των Βάσκων. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχει πρόβλημα ε, διαμεθοριακής διακυβέρνησης το οποίο προκύπτει και από την πρόταση που μας έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ένα συντονιστή ο οποίος αντί να βελτιώσει τα πράγματα τα επιδίνωσε. Έγιναν τα πράγματα ακόμα πιο δύσκολα και αυτή τη στιγμή στα μισά της διαδρομής ε, μας προτείνεται μια πλήρη αλλαγή των κανόνων. Θα ήθελα να μας πείτε με ποιο τρόπο θα καταφέρουμε να βελτιώσουμε όλα όσα θέλαμε να επιτύχουμε στι δημοσιονομικέ προπτικές. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μπιλμπάου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον Επίτροπο για τις εξηγήσεις που μας έδωσε. Σήμερα το πρωί είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε τους υπεύθυνους ε, για τα θέματα του προπολογισμού και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο Σέτσι για τα όσα έκανε για τη γραμμή προπολογισμού 3. Μετά όμω από τη σημερινή συνεδρίαση θα ήθελα να σα θέσω την εξή ερώτηση. Εσεί, σε αυτή την τροποποίηση των κριτηρίων ε, με βάση τι νέε δημοσιονομικέ προπτικές αναφερθήκατε στα διευρωπαϊκά προβλήματα. Το ε, ε, ε, Βάσκαο, το πρόγραμμα για τη χώρα των Βάσκων, έχει σοβαρό διαμεθοριακό πρόβλημα. Επίση, υπάρχει πρόβλημα στην εκτέλεση τη γραμμή προπολογισμού 3 φέτο και δημιουργείται πρόβλημα και με τη γαλλική πλευρά και με τη γαλλική κυβέρνηση διότι ε, υπάρχουν δυσκολίες στην επίλυση του θέματος. Θα ήθελα να ρωτήσω λοιπόν αν η γραμμή προπολογισμού 3 βρίσκεται μεταξύ των κριτηρίων που θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε προκειμένου αυτή η γραμμή προπολογισμού ε, να εξοποιηθεί και να ε, κατά πόσον ελοχεύει ο κίνδυνο να μείνει χωρί πόρου. Θα ήθελα να σας παρακαλώ να μου απαντήσετε σε αυτή την ερώτηση. Η κυρία Ράνερα για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πίτροπε για την ε, παρουσίασή σας αυτή. Δεν ε, θα ε, κάνει σε κανένα εντύπωση αν ε, αναφερθώ στο τούνελ Μπρέμερ. Ε, ήδη αναφέρθηκε ο συνάδελφος αυτό. Η ερώτησή μου κύριε Πίτροπε είναι μπορείτε να πείτε ήδη τώρα τι μέτρα προβλέπετε αν ε, δεν δεσμευτούν η Αυστρία και η Γερμανία όσον αφορά το ξεκίνημα του έργου. Ε, ευχαριστώ κύριε Ράνερ. Ο κύριος Λάιχτφριντ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν ε, όσον αφορά τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Νομίζω ότι έχουμε δύο δυνατότητες και θα πρέπει να αποφασίσουμε. Θέλουμε χρηματοδότηση διευρωπαϊκών δικτύων στο μέλλον που να ε, χρηματοδοτεί του εθνικού ή του διεθνεί ε, διαδρόμου. Δεν νομίζω ότι έχουμε αρκετά χρήματα για να κάνουμε και τα δύο. Και πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει περισσότερο την, ε, το καθήκον να χρηματοδοτεί διασυνοριακέ συνδέσει. Και δεύτερον, θέλουμε πάλι ένα ωραίο δίκτυο που να λαμβάνουμε υπόψη όλα τα απαραίτητα ή θέλουμε πραγματικά να γίνει κάτι για, τα, για τους κυρίως, ε, για τις ε, ναυτιλιακές ε, μεταφορές. Θα πρέπει λοιπόν να ποντάρουμε εκεί όπου τα κράτη-μέλη είναι διευθυμένα να κάνουν κάτι και να συγχρηματοδοτήσουν, γιατί αλλιώ δεν θα κάνουμε τίποτα στο τέλο. Είναι σημαντικό τα δύο αυτά θέματα, θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μα κατά τον προγραμματισμό νέων δικτύων και διαδρομών άλλο. Ε, χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω το, ε, το θέμα των ε, τελών στα αεροδρόμια, αλλά δεν γίνεται τίποτα και αυτό είναι κακό. Ε, μιλάμε για ε, διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κανένας όμως δεν συζητάει πώς θα χρηματοδοτηθούν όλα αυτά. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω τι σχεδιάζετε συγκεκριμένα, ώστε το Συμβούλιο που δεν έχει κάνει τίποτα, να αναγκαστεί να λάβει κάποια απόφαση και να προχωρήσει. Ευχαριστώ κύριε Λάιχτφριντ. Ο κύριο Τουμόλ, σαν δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλώ όρισατε κύριε Κάλλα στην Επιτροπή μα και σας ε, συγχαίρω για τι εργασίε σα. Πολύ σύντομα. Βρισκόμαστε σε ένα πλαίσιο οικονομική κρίσεω και δεν θα μπορέσουμε να έχουμε πόρου για όλα τα προγράμματα. Αυτό που θα ήταν ενδιαφέρον να γνωρίζουμε από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ποιες ε, θα είναι οι αναλύσεις οικονομικών επιπτώσεων προκειμένου να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι θα υλοποιηθούν τα προγράμματα που έχουν μεγαλύτερη μακροοικονομική ανάπτυξη για την ευρωπαϊκή οικονομία. Για μένα αυτό είναι σημαντικό πρέπει να υπάρχει μια κάποια βαθμολόγηση, μια κάποια αξιολόγηση, ανάλυση κόστους ωφελίας για τις μακροοικονομικές επιπτώσεις, για τα ωφέλη ε, σε όρους οικονομικής ανάπτυξης που θα μπορούσαν να επιφέρουν τα διάφορα προγράμματα για την ευρωπαϊκή οικονομία. Διότι ε, δεν μπορούμε να έχουμε την πολυτέλεια να μην λάβουμε υπόψη ε, κριτήρια που αφορούν την οικονομική αποτελεσματικότητα σε περίοδο κρίσης. Εγώ προέρχομαι από την Ισπανία, η οποία για 20 χρόνια ελάμβανε χρηματοδότηση από το Ταμείο συνοχή και τα περισσότερα προγράμματα υλοποιήθηκαν χωρί τη χρήση κριτηρίων οικονομική ανάπτυξη. Στη συνέχεια είχαμε μια πολύ σημαντική οικονομική κρίση και φαίνεται ότι υπάρχουν αποκλήσει μεταξύ χωρών Δύσης και ε, Νότου και Βορρά, διότι λάμβαναν χρηματοδότηση για πολλά χρόνια, αλλά δεν ε, ακολουθούσαν κριτήρια οικονομική αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητας. Ε, νομίζω ότι και η ώρα να αλλάξουν τα πράγματα. Ευχαριστώ κυρία Λίχτεμπεργκερ για δύο λεπτά. Θα ήθελα να επανέλθω στην, ε, στην προσούρα, ε, στο έγγραφο αυτό. Ε, είναι πολύ καλή η αποτίμηση αυτή και θα μπορεί να αποτελεί πολύ καλή βάση, αλλά κάτι λείπει. Θα πρέπει, όπως προβλέπεται στο ευρωπαϊκό δίκαιο, τα σχέδια αυτά να αποτελέσουν αντικείμενο περιβαλλοντικής μελέτης. Και δεύτερον, όσον αφορά τη χρηματοδότηση από τα κράτη-μέλη. Ε, δεν θα κάνουμε αποκλειστική χρηματοδότηση κανενός προγράμματος, ε, αλλά οι διαφορετικές προϋποθέσεις στα παλιά και νέα κράτη-μέλη, διότι στα νέα μπορεί να υπάρξει χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής. Ε, αυτό δεν μπορεί να γίνει στα παλιά κράτη-μέλη και αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα μεγάλα έργα, Γερμανία, Αυστρία, Ιταλία, που δεν μπορούν να ζητήσουν τέτοια χρήματα. Και η Αυστρία αν πει τώρα ότι επειδή από την Ιταλία δεν έχουμε σαφή απάντηση σχετικά με την παράταση των ε, σιδηρομικών ε, δικτύων, ε, μπορούμε να μεταφέρουμε το βάρος στους φορολογούμενους και να πούμε ότι θα περιμένουμε να δούμε αν θα λάβουμε μια καλή απάντηση. Έτσι, όσον αφορά την διετία που αναφέρεται στα πολύ μεγάλα αυτά έργα, μήπως θα πρέπει να δώσουμε περισσότερο από δύο χρόνια παράταση και αν ναι, μήπως ε, θα πρέπει να εξετάσουμε τη δυνατότητα να επιτρέψουμε ε, εναλλακτικά προγράμματα τα οποία να είναι πιο οικονομικά. Αυτό θα ήταν σημαντικό για μένα και Ε, και επίση, όσον αφορά τις, ε, τα έργα Aeronel και τη διασύνδεση ε, Βρυξελών-Στρασβούργου, αυτά έχουν πολύ, καλή, πολύ κακή βαθμολογία στην έκθεση αυτή. Μπορείτε να μου το εξηγήσετε αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Βούλης. Έχω μια συγκεκριμένη ερώτηση προς εσάς κύριε πίτροπε. δεν με ακούτε όμως. Θα ξεκινήσω από την αρχή. Σας παρακαλώ να με ακούσετε, δύο λεπτά έχω. Έχω μια συγκεκριμένη ε, ερώτηση κύριε Κάλλας. Ε, το πρόγραμμα 20 στο έγγραφο που μας δώσατε, στην προσούρα που μας δώσατε, ε, είναι μια σύνδεση με πλοίο και αναφερόμαστε στην διαδρομή Λούιμπεκ-Πούτγκαρντεν. Ε, η νήσος ε, Φέμαν ε, απειλείται διότι πέρα από τη συνδρομική γραμμή θα χτιστεί και δρόμος. Εγώ είμαι από το Αμβούργο και αυτό είναι πρόβλημα και για το Αμβούργο εάν έχουμε περισσότερα φορτηγά στη διαδρομή αυτή. Υπάρχει μια πρωτοβουλία κατά της σταθερής αυτής σύνδεσης και η ερώτησή μου είναι κατά πόσο λαμβάνετε αυτό υπόψη από εσά και ε, εάν ε, έχει δοθεί θετική απάντηση και αν μπορεί να πραγματοποιηθεί ε, ένα τέτοιο έργο τη στιγμή που δεν υπάρχουν χρήματα και που υπάρχει μια πολύ καλή σύνδεση με φεριμπότ για τα ε, αυτοκίνητα και τα φορτηγά. Ε, θα πρέπει να γίνει και περιβαλλοντική μελέτη για να εξεταστούν οι επιπτώσεις ε, στη θάλασσα και στο υπόλοιπο περιβάλλον. Θα ήθελα να το αναφέρω αυτό διότι θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό θέμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Στέρξ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Θα ακούσω με μεγάλη προσοχή τις απαντήσεις που θα δώσει η κυρία Ρίχτεμπέργκερ για τη σιδηροδρομική γραμμή του Ρήνου. Μία δεύτερη ερώτηση. Λέμε ότι η προθεσμία είναι το τέλος του 2015. Ενδεχομένως, ορισμένα ενδιαφέροντα έργα θα πρέπει να έχουν κάποια προτεραιότητα. Αναφέρομαι σε αυτό τη Σκέλντα. Ένα τέτοιο πρόγραμμα ενδεχομένως θα έβαζε τέλος σε μια δύσκολη οικονομική κατάσταση. Η, τελική, καταληκτική ημερομηνία του 2015 είναι απόλυτη ή θα ληφθούν υπόψη διάφορα στοιχεία που θα μπορούσαν να, να οδηγήσουν σε μια τροποποίηση ημερομηνία. Μιλάμε για 44 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά δεν ξέρουμε από πού θα πρέπει να γίνει αυτή η αποταμίευση. Κύριε Κάλλας, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας όσον αφορά αυτά που θα πρεπει να γινει αυτη η αποταμιευση κυριε σε συμφωνω απολυτα μαζι σας οσον αφορα αυτα που προτεινετε στην έκθεση αυτή ε, και όσον αφορά την χρηματοδότηση. Ε, δεν θα πρέπει να αλλάξουμε τους κανόνες ε, του παιχνιδιού στη μέση του παιχνιδιού. αλλά τουλάχιστον έχουμε έναν επίτροπο που παίρνει στα σοβαρά τους ε, κανόνες του παιχνιδιού. Αναφερθήκατε σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και λαμβάνετε υπόψη σα ότι δεν μπορούν όλα τα προγράμματα να ολοκληρωθούν. Μπορεί λοιπόν να δοθεί παράταση διετίας. Δεν ε, σταματάει η Ευρωπαϊκή Ένωση τα προγράμματα, τα κράτη-μέλη τα σταματάνε. Ε, εφόσον δεν ε, τα εφαρμόζουν σωστά και δεν ε, προσπαθούν να βρουν τις ιδανικέ λύσεις ακούγοντα και τι έχουν να πούνε οι κάτοικοι. Πρέπει λοιπόν συγκεκριμένα τα κράτη-μέλη να κάνουν κάποια πράγματα, διότι αλλιώς διακυβεύονται τα έργα. Στην κυρία Ρίλτε να πω ένα πράγμα. Δεν υπάρχει στο ε, βιβλίο αυτό ένα έργο ε, για το οποίο να μην ε, λαμβάνει θυμωμένα γράμματα ο Επίτροπος από τους κατοίκους. Θα πρέπει λοιπόν εγκαίρως να έρχονται σε επαφή τα κράτη-μέλη με τους κατοίκους για να βρουν τις βέλτιστες λύσεις. Ευχαριστώ κύριε Σκούν, δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για την λεπτομερή παρουσίαση Ε, και που μένεται στην στρατηγική 20.002 την οποία μαζί έχουμε καθορίσει. Μιλάμε για μεταφορά των μεταφορών από, τον, από τις οδικές ε, μεταφορές στη θάλασσα και στους σιδηροδρόμους. Και ακούσαμε πολλούς ε, ομιλητές από την Γερμανία η Γερμανία όμως είναι η μεγαλύτερη, ο μεγαλύτερος χώρος διέλευσης στην Ευρώπη. Αν θέλουμε να συνδέσουμε τις διάφορες περιφέρειες της Ευρώπης, αυτό επηρεάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό την Γερμανία. Ε, γι' αυτό το θέμα επηρεάζει περισσότερο από εμά και γι' αυτό θα πρέπει ε, πολύ προσεκτικά να εξετάσουμε το θέμα. Η ε, πρωτοβουλία της Βελγικής Προεδρίας είναι αξιέπαινη για μεγάλα φορτηγά να ε, έχουμε διόδια, να έχουμε κάποια τέλη. Στη Γερμανία αυτό το κάνουμε εδώ και πολύ καιρό, αλλά κύριε Επίτροπε, ίσως θα πρέπει να έρθετε σε επαφή με τους συναδέλφους σας και να πείτε ότι τα χρήματα που ε, συλλέγονται στο μέτρο μεταφορών από ε, τα διόδια, ε, από τα διάφορα τέλη, να διατίθενται πάλι στον χώρο των μεταφορών, ιδιαίτερα για τα, τους ευρωπαϊκούς άξονες. Ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε όλους τους 18 ομιλητές. Έχετε λοιπόν υλικό για να μας απαντήσετε. Κύριε Επίτροπε, έχετε 10 με 11 λεπτά. Παρακαλώ. Thank you very much. Uh, all... Ευχαριστώ. Σαφέστατες οι απαντήσεις, οι ερωτήσεις σας. Θέσατε πάρα πολλά θέματα. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όσο γίνεται περισσότερες από τις ερωτήσεις που ετέθησαν. Ένα σημαντικό θέμα ετέθη από τον κύριο Αλχαντράουι. Τι θα συμβεί με αυτά τα κονδύλια και ποιες θα είναι οι προτεραιότητες για την ανακατανομή αυτών των 311 εκατομμυρίων. Υπάρχουν δύο ιδέες. Η πρώτη ιδέα είναι, βεβαίω πρόκειται για ένα μικρό χρηματικό ποσό, λαμβάνοντα υπόψη το μέγεθο των έργων αυτών. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε προ δύο κατευθύνσει. Μία ιδέα είναι να ετοιμαστούμε για τις ε, επόμενες δημοσιονομικές ε, προοπτικές. Η δεύτερη ιδέα είναι να χρηματοδοτήσουμε μικρά κομμάτια του έργου. Θα μπορούσαμε να χρηματοδοτήσουμε ε, κάτι σε κάποιο άλλο τομέα. Ας πούμε κάτι που να έχει σχέση με την τεχνολογία του TNT. Αυτές είναι μερικές προκατακτικές ιδέες. Βεβαίως δεν έχουμε καθορίσει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο που να μπορεί να εφαρμοστεί από όλους τους δικαιούχους. Το ερώτημα το άλλο είναι ποια είναι η σχέση με τις επόμενες δημοσιονομικές ε, προοπτικές. Ποιες είναι οι σχέσεις αυτών των περικοπών. Δεν είναι μπορούμε να πούμε ότι όλα αυτά δεν μπορούν να εφαρμοστούν και πάλι. Θα πρέπει όμως να γίνει μία επαναξιολόγηση. Δηλαδή δεν θα πρέπει να δοθεί εντύπωση ότι θα κάνουμε περικοπές από το 2015 αλλά ενδεχομένω θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε. Όχι, δεν δίνουμε αυτές τις υποσχέσεις, αυτό είναι ένα καινούριο έργο και θα πρέπει να συζητηθεί ως τέτοιο. Το ενδιαφέρον ερώτημα είναι είναι συνετό το να γίνουν αυτές οι περικοπές. Υπάρχουν ε, ορισμένοι που ζητάνε περισσότερα κονδύλια. Ε, ο συνάδελφός μου, Μούλερ, είναι υπεύθυνο για θέματα απαλλαγής. Ε, η δική του άποψη είναι ότι πρέπει να γίνουν περικοπές αν δεν χρησιμοποιούνται τα χρήματα. Ετέθη ένα θέμα από πολλά από τα μέλη του Κοινοβουλίου και αυτό σε σχέση με τα μεγάλα προγράμματα ή την προπαρασκευαστική διαδικασία ε, που έχει σχέση με τις ε, επιδράσεις στο περιβάλλον. Το τρομερό είναι ότι Έχουμε έναν κατάλογο, αυτός ο κατάλογος έχει αυξήσει το κόστος και αυτό είναι ένα δίλημα για όλους τους συμμετέχοντες καταρχάς για τις χώρες μέλη. Τα προβλήματα ξεκινάνε με την έναρξη του έργου έχουν γίνει λοιπόν οι αξιολογήσεις, έχουν, γίνει, έχουν ληφθεί οι άδειε και ε, ε, αρχίζει η εφαρμογή. Και εκεί ξεκινάνε και οι συγκρούσεις. Καταλαβαίνετε ότι αυτή δεν είναι μια πολύ καλή κατάσταση για το επόμενο TNT. Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι ότι θα πρέπει να σκεφτούμε ε, αν προγραμματίζουμε χτίζουμε καινούρια στοιχεία υποδομών, τα οποία θα μπορούσαν να δημιουργήσουν πολλές αντιρρήσεις ή επικεντρωνόμαστε στην ανάπτυξη των υπαρχόντων δικτύων, στην ε, ανανέωση ε, των ε, κτηρίων, στην αύξηση του δυναμικού της χωρητικότητας. Θα έλεγα όμως ότι η διαδικασία αυτή είναι ιδιαίτερα διαφανής ε. και εμείς προσπαθούμε να συζητήσουμε με όλους τους ενδιαφερόμενους, με μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με προσώπους ε, της κοινωνίας των πολιτών, των χωρών μελών, για να προβλέψουμε όλα αυτά τα προβλήματα που θα μπορούσαν να ανακύψουν και για να αποφύγουμε ξαφνικά να έχουμε ένα έργο και να χρειαστεί να το διακόψουμε γιατί προέκυψε κάτι απρόοπτο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα ταμεία συνοχής και τη σχέση μεταξύ των ταμείων συνοχής, φαντάζομαι ότι η Γενική Διεύθυνση Ρέτζο έδωσε περίπου 20 δις που χρησιμοποιούνται ε, για τις μεταφορές. Είναι από το ε, Ταμείο Συνοχής. Ε, ε, εκείνο που μπορώ να πω είναι ότι σε συνεργασία με τον Επίτροπο Χάν προσπαθούμε να συντονίσουμε τις πολιτικές και να επιτύχουμε μια καλύτερη συνοχή. Εναπόκειται βέβαια στις χώρες μέλη που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι για τα διάφορα θέματα. αρκετά θέματα αφορούσαν ένα μεγάλο ε, έργο, τον Μπρένερο. Ο Πατ Κόξ ε, που είναι ο συντονιστής ε, για αυτό το PP 1 θα έρθει και θα μπορέσει να απαντήσει αργότερα στις ερωτήσεις σας. Δεν σημαίνει όμως ότι όλα τα έργα είναι τα ίδια. Ελπίζω ότι με αυτά τα οκτώ δις αυξήσουμε τη χρηματοδότηση του επόμενου TNT. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για ένα μικρό χρηματικό ποσό. Εμείς μιλάμε για 500 δις για να αναπτυχθεί όλο το δίκτυο. Ενδεχομένως είναι πάρα πολλά, αλλά δεν θα προέρχονται ποτέ από το ευρωπολογισμό. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει ένας συνδυασμός όλων των πόρων, εάν θέλουμε να αναπτύξουμε τις υποδομές. Και ο προπολογισμό μπορεί να δώσει ορισμένα κονδύλια, ορισμένα ε, στοιχεία ε, κομβικά. Και εμεί θα πρέπει να τα εντοπίσουμε αυτά. Θα προσπαθήσουμε βεβαίως να μην τα μπλοκάρουμε τα χρήματά μας σε μεγάλα έργα που σε κάθε περίπτωση θα διακοπούν. Αυτά σε ό,τι αφορά τα μεγάλα έργα. Κάτι άλλο που αφορά το θέμα της χρηματοδότησης. Συζητήσαμε πολλές φορές για το πώς θα μπορούσε να βρεθεί επιπρόσθετη χρηματοδότηση. Εγώ συναντήθηκα με πάρα πολλού ιδιωτικού επενδυτέ με επενδυτικές τράπεζες, με την Goldman Sachs, με την Macquarie και μου υπέβαλαν πολύ ενδιαφέρουσε προτάσεις. Το θέμα είναι ότι όλα αυτά θα πρέπει να είναι μακροπρόθεσμα. Δεν θα πρέπει να παρεμβαίνετε και δεν θα πρέπει ε, να υπάρχουν πολιτικές διακυμάνσεις. Εκείνο που μου είπαν είναι ότι η βασική ιδέα είναι ότι είναι καλύτερα να ανανεώνουμε υπάρχοντα δίκτυα. Διαφορετικά θα πρέπει να αγοράσουμε ε, τη γη, τα οικόπεδα που είναι βεβαίως πάρα πολύ ακριβά. Το ό,τι αφορά το έργο της ε, Βαλτικής Η κυβέρνηση της Λιθουανίας αποφάσισε να επανεξετάσει την όλη δομή του έργου έτσι ώστε θα είναι λιγότερο δαπανηρό. Πολύ θετική αυτή η απόφαση. Πιστεύω ότι η κυβέρνηση της Λιθουανίας δήλωσε ότι έχει αποφασίσει προς, προς τα που θα εξελιχθεί το σιδηροδρομικό της ε, δίκτυο. Πολύ σημαντικό αυτό για το σιδηροδρομικό δίκτυο της Βαλτικής. Ε, αυτό είναι ένα δίκτυο εμπορευμάτων. Αν θέλουμε να αναπτύξουμε το δίκτυο επιβατών θα πρέπει να σκεφτούμε μία σύνδεση βορρά-νότου. Αλλά βεβαίως πολλά εξαρτώνται από τη δέσμευση των ε, ενδιαφερομένων κυβερνήσεων. Η Λιθουανία επίσης αποφάσισε να αναπτύξει αναπτύξει το συνδρομικό της δίκτυο και τώρα έχουμε την Εστονία και την λετονία που θα πρέπει επιτέλους να αποφασίσουν. Φαντάζομαι ότι οι συντονιστές μπορεί να σχολιάσουν συγκεκριμένα ε, προγράμματα στο ε, στην προτεραιότητα 3 δεν θα υπάρξουν ε, περικοπές. Οι ε, εσωτερικές πλωτοί οδοί είναι όντως ένα πρόβλημα και πραγματικά εκεί είμαστε αρκετά απεσιόδοξοι για την σύνδεση δηλαδή Ρήνου και Δούναβη. Θα πρέπει να συνεργαστούμε με τους συντονιστές με τον κύριο Σέλτες και την κυρία Μπέισης. Αλλά θα πρέπει να συνεργαστούμε και με τις κυβερνήσεις. Έχουμε λοιπόν πολλή δουλειά να κάνουμε με τις κυβερνήσεις. Πολλά εξαρτώνται από τις κυβερνήσεις και από τη δική μου την πλευρά θα ήθελα να διευκολύνω τη συνεργασία μεταξύ των κυβερνήσεων. Βεβαίως ε, μπροστά μας έχουμε δύσκολο δρόμο γιατί πολλά έργα εξαρτώνται από 10 ε, χώρες. Όταν έχουμε να κάνουμε με δύο χώρες τα πράγματα είναι ευκολότερα. Εδώ τα πάντα εξαρτώνται από τη συνεργασία. Μέχρι στιγμής καλά πήγαν τα πράγματα. Αρκετά έχουν γίνει στο TNT και βεβαίω μπορούμε να επικρίνουμε ορισμένα πράγματα. Μακάρι να μπορούσε να υπάρχει μια καλύτερη διασύνδεση μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα πολύ σημαντικό ε, έργο για την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς. Ευχαριστώ πολύ. Στην ώρα μου τελείωσε, λέει ο Επίτροπος. Σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας. και είμαστε στην ώρα μας. Ελπίζω να μπορέσουμε να κρατήσουμε αυτή την καλή συνήθεια και για το υπόλοιπο απόγευμα. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ και προσβλέπουμε στην επόμενη συνάντησή μας. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ, εξέλχεστε ησύχως. Get Για να συνεχίσουμε. Να ζητήσω από τους συντονιστές να έρθουν εδώ στο Προεδρείο Uh, Ωραία. Θα παρακαλούσα τους ε, κυρίους Κότς, Μπάλας, Μπρίνκορτ, Βίνκ Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, για περάστε για να τηρήσουμε λίγο και το χρονοδιάγραμμα. Περνάμε στο επόμενο σημείο λοιπόν της ημερήσιας διάταξης. Σας παρακαλώ τα πηγαδάκια να περάσουν έξω, σας παρακαλώ, αν γίνεται διότι η μόνη συνεδρίαση που έχει σημασία είναι η δική μας. Ωραία λοιπόν. Σημείο 13 στην διάταξη, ανταλλαγή απόψεων με τους συντονιστές, τους υπόλοιπους συντονιστές και για να εξηγήσουμε λίγο στους συναδέλφους τι κάναμε σήμερα το πρωί. Θα ήθελα ο καθένας από εσά να κάνει μια εισογωγή 10 λεπτών ο ένας μετά τον άλλον. Στη συνέχεια θα έχουμε ερωτήσεις και σχόλια από τα μέλη και κατόπιν θα σας ζητήσω εάν υπάρχει χρόνος να απαντήσετε ο, ένας, ο καθένας με τη σειρά του όπως ε, και στην αρχή. Αυτό για να είμαστε βέβαιοι ότι θα έχουν τη δυνατότητα να μιλήσουν και όλα τα μέλη και όχι μόνο οι συντονιστές. Ε, θα ξεκινήσω λοιπόν με τον κύριο Κόξ, ο οποίος ε, έχει το πρόγραμμα προτεραιότητας περιθμών 1. Ο ΠΑΤ είναι ένα ακόμα μέλλον ε, της ομάδας των παλιών φίλων του Κοινοβουλίου. Είχαμε μια συνάντηση παλιών φίλων, είδαμε κάποιους και το πρωί, τώρα εσένα. Έχεις το χρόνο λοιπόν το λόγο για 10 λεπτά. Κύριε, Κύριε Πρόεδρε, Κύριοι βουλευτές, χαίρομαι ιδιαίτερα που επιστρέφω εδώ. Είναι η πρώτη φορά που επανέρχομαι μετά από την ακρόαση πριν από μερικούς μήνες. Προσπάθησα να αναπτύξω κάποιο ρυθμό σε αυτό το ε, σε ό,τι αφορά αυτό το θέμα. Θα βρείτε τι λεπτομέρειε στην ετήσια έκθεση σε κάθε περίπτωση. Εάν θα έπρεπε να ανακεφαλαιώσω τρία θέματα που θα επιθυμούσαν να συμβούν και όπου θα εστιατεί η προσοχή μου είναι το να αναφερθούμε σε συγκεκριμένες δεσμεύσεις για το ξεκίνημα της ε, ε, φάσης 3 ε, στη σύραγγα του Μπρένερο. Δεύτερον, να προωθήσουμε την ιδέα της απαραίτητης το πόσο απαραίτητο είναι να, αναπτυχθούν, να αναπτυχθεί ο άξονα βορρά νότο και τρίτον το να δοθεί προτεραιότητα στην εξέλιξη της, στην ανάπτυξη της συζήτησης σχετικά με τα συνοδευτικά μέτρα έτσι ώστε να όταν υπάρχει, όταν θα υπάρξει η απαραίτητη υποδομή να μπορέσουμε να κινηθούμε. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Αυστρία. Είναι ένα θέμα στο οποίο αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία. Σε ό,τι αφορά το δικό μου ρόλο, είπα ότι ο ρόλος της ακρόασης είναι η συνεργασία και η διαβούλευση. Πιστεύω ότι σε ό,τι αφορά τα μεγάλα αυτά προγράμματα υποδομών, ένα θέμα που έχει θυγεί αρκετέ φορέ τον Επίτροπο σήμερα τα απόγευμα. Πιστεύω λοιπόν ότι δίνεται μεγάλη σημασία στην αξιολόγηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον σε θέματα που αφορούν τον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό. Επίσης, προσπαθούμε να δούμε τι είναι αυτά τα μακροχρόνια προγράμματα και προσπαθούμε αυτό να το ε, μεταφέρουμε και προς τα έξω. Εκεί νομίζω ότι υπάρχει ένα ε, πρόγραμμα. Το PP1, e όπως γνωρίζετε, είναι ένα, είναι βαρχίδα θα λέγαμε των ε, προτεραιοτήτων. Υπάρχει το 95% των κονδυλίων για το 10 Πολλά έχουν γίνει από τον προκάτοχό μου, τον Κάρεν Βαν Μίτ και εγώ βέβαια εποφελούμε. Έγινε μια δήλωση το 2009 στη Ρώμη. Αυτό οδήγησε στην παράδοση και στην ουσία αυτό με ενδιαφέρει. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε κάτι αυτό. Στις 19 Νοεμβρίου, σε λίγες εβδομάδες δηλαδή, θα έχω τη χαρά για πρώτη φορά να παραστώ σε μια διακυβερνητική συνάντηση μεταξύ της Αυστρίας και της Ιταλίας. Επιτρέψα μου να επανέλθω στο θέμα αυτό σε λίγο. Και στις 13 Νοεμβρίου ελπίζω να συναντηθώ με τους προέδρους των ομάδων εργασία, οι οποίοι προεδρεύουν διαφόρων ομάδων εργασίας ε, σε μια προσπάθεια να κατανοήσω τι ακριβώς γίνεται για να εντοπίσω τι δεν έχει γίνει αλλά και για να θέσω στόχους για το τι πρέπει να γίνει και για να μπορέσω λεπτομερέστερα να αναφερθώ σε αυτά τα θέματα ενώπιόν σας στο μέλλον. Η ετήσια έκθεση αναφέρει λεπτομερώς τι έχει συμβεί σε ό,τι αφορά το PP1 αρκετά καλά πράγματα έχουν συμβεί στη Γερμανία, καλά έχουν συμβεί στην Αυστρία και καλά έχουν συμβεί και στην Ιταλία. Όπως όλα αυτά τα προγράμματα, το υλικό που λείπει είναι τα καλά πράγματα που συμβαίνουν και που συνδέουν όλα τα υπόλοιπα σε μια ευρωπαϊκή βάση. Συνεπώς, κατά κάποιο τρόπο έχουμε μια επιβεβαίωση σε αυτό το έργο Ναυαρχίδα, όπως σας το περιέγραπα. Ε, η Επιτροπή αναφέρθηκε σε ένα πάσχο, σε ένα ψηφιδωτό δικτύων έγινε κάποια παρέκκληση από τις προθεσμίες. Θεωρήσαμε ότι η πρώτη διό... Ε, σύραγγα το βράδυ ήταν έτοιμη φέτος, πράγμα που δεν έγινε. Επιτρέψτε μου να πω ότι έχω την αίσθηση και αυτό προέκυψε από τις ερωτήσεις και τις παρατηρήσεις σας, ότι ως ένα βαθμό ε, είχαμε να κάνουμε με μια λογική αν η κότα έκανε τα αυγό ή το αυγό την κότα μεταξύ των βασικών συντελεστών η μία ομάδα κοιτάει την άλλη στην άλλη πλευρά των σύνορων και να λένε αν εσείς κάνετε αυτό θα κάνουμε και εμείς το άλλο. Και οι άλλοι κάνουν ακριβώς το, το ίδιο. Το πρόβλημα με τη λογική της κότας και του αυγού είναι ότι δεν ξέρετε πότε θα οδηγηθεί σε μια πραγματική δέσμευση γιατί είναι ένα κυκλικό θεώρημα, μια κυκλική λογική. Λοιπόν θα πρέπει να μεταφερθούμε από την κότα και το αυγό στο αυγό και το μπέικον. Να σας εξηγήσω. Το μπέικον και το αυγό ε, έχει την, ε, ε, είναι κάτι το οποίο έχει απόλυτη δέσμευση, έχει τη δέσμευση του χοιρινού από το οποίο παράγεται. Θα πρέπει λοιπόν να ενθαρρύνουμε με έναν σταθέστατο τρόπο μία δέσμευση έτσι ώστε το 2011 θα ξεκινήσουμε με βάση δύο στοιχεία στη Σύρια και Σύρια του Μπρένου από δύο πλευρές, από την Αυστρία και από την Ιταλία. Και είναι προσδοκία και πεποίθησή μου κύριε Πρόεδρε ότι αυτό είναι στα όρια του εφικτού. Αυτό που συμβαίνει και στην Ιταλία και στην Αυστρία και άκουσα μερικά από τα σχόλια που διατυπώθηκαν προηγουμένως ενώπιον του Επιτρόπου ότι η προσοχή εστιάστηκε σε αυτό που λέμε κατασκευή. Δηλαδή, αλλά σε κομμάτια, σε τμήματα. Μία κατατμήματα αντιμετώπιση. Δηλαδή, μερικές φορές μπλοκάρεται όλο το έργο γιατί δεν μπορεί κανείς να το αντιμετωπίσει σταδιακά και σε κομμάτια. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει, να ληφθεί μία απόφαση και από τις και θα πρέπει να βρεθούν και τα κονδύλια να εντοπιστούν σε αυτή τη φάση. Κύριε Πρόεδρε, η άποψή μου λοιπόν είναι ότι κινούμεθα προς κάτι απτό, πραγματικό, οριστικό. Προσπαθούμε δηλαδή να ξεφύγουμε από αυτή τη λογική της κότας και του αυγού και να φτάσουμε στη λογική του μπέικον και του αυγού. Αν τα καταφέρουμε νομίζω ότι ε, αυτό θα γίνει τον επόμενο χρόνο. Εάν συμβεί πραγματικά θα έχουμε επιτελέσει σημαντική πρόοδο. Δεν είναι βεβαίω σίγουρο. Εσείς έχετε μεγαλύτερη πείρα από μένα με τον Υπουργό τι όλοι και τους αξιωματικούς του Υπουργείου στη Ρώμη, με τον Υπουργό Μπούντα στη Βιέννη και με τον Υπουργό Ράμσαν και τους ε, συνεργάτες του στο Βερολίνο παρόλες τις οικονομικές ε, πιέσεις, παρόλο το πρόγραμμα εθνικής αναθεώρησης θα υπάρξει μια σοβαρή δέσμευση έτσι ώστε να τεθούν τα θέματα επιτάπητος και να υπάρξουν κονδύλια για τα ξεχωριστά κομμάτια του έργου. Θα τεθεί το θέμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όλοι θέλουν να γνωρίζουν τι θα σημαίνει αυτό για την ευρωπαϊκή πλευρά αυτή τη εξίσωσης και πιστεύω ότι αυτό ισχύει για οποιοδήποτε έργο εξετάζεται. Thank you very much, Mr. Cox. Ευχαριστώ κύριε Κόξ. Ο κύριος Μπάλα στη συνέχεια, ο οποίος είναι υπεύθυνο για το πρόγραμμα προτεραιότητας 17 ένα που ενδιαφέρει ιδιαίτερα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διότι είναι αυτό το οποίο περιλαμβάνει το Στρασβούργο. Κύριε Μπάλατ. Um, uh, uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το πρόγραμμά μου είναι το 17, που είναι ε, Ανατολή Δύση, Παρίσι, Μπαρατισλάβα. Πρόκειται για μια διεθνή γραμμή που διασχίζει και κάποιες άλλες γραμμές προτεραιότητας σε σημαντικούς κόμβους και ίσω το πιο σημαντικό σημείο συνάντησης είναι με το πρόγραμμα προτεραιότητας 1 στο Μόναχο όπου φαίνεται ότι επικεντρώνονται οι περισσότεροι σιδηρόδρομοι. Ένα από τους κόμβους συνάντησης είναι αυτός περιλαμβάνονται αρκετά ε, για τρει από αυτές ε, έχουμε την πρωτεύουσα στη γραμμή και σε δύο αυτή είναι η κύρια πρόσβαση για την ίδια την πρωτεύουσα. Αυτό συμβαίνει στην Αυστρία και στη Σλοβακία. Η Βιέννη και η Μπρατισλάβα θεωρούν ότι αυτή η γραμμή είναι ιδιαίτερο σημαντική. Για το Παρίσι η σημασία της γραμμής ε, είναι αναδυόμενη Αν το δείτε από το Παρίσι είναι το TGV Est, το νέο άνοιγμα προς τις αναδεόμενες αγορές. Στη Γερμανία η κατάσταση είναι λίγο διαφορετική γιατί η συγκεκριμένη γραμμή απέχει ε, μεγάλη απόσταση από το Βερολίνο, βρίσκεται στο βαθύ νότο αν θέλετε της Γερμανίας και είναι σημαντική ε, από οικονομικής πλευράς ε, και οι συνδέσεις ε, και από τις δύο πλευρές θα πρέπει να επισημαίνονται. Θα πρέπει να πω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι γίνεται καλή πρόοδος για τη συγκεκριμένη γραμμή. Περίπου το 40% έχει ολοκληρωθεί και άνω του 20% είναι να εξελίξη, που δεν είναι και πολύ άσχημο αποτέλεσμα αν λάβουμε υπόψη ότι θα πρέπει να τηρούμε τις προθεσμίες και τις ημερομηνίες στόχους να σας αναφέρω κάποια από τα καλά μας αποτελέσματα. Υπάρχει άμεση σύνδεση με σιδηρόδρομο μεταξύ Γερμανίας και Γαλλίας, μεταξύ Στουτγκάρδης μέσω της Καρλούε στη Παρίσι. Και από τότε που ξεκίνησε η λειτουργία αυτής της γραμμής, πριν από τρία χρόνια, περίπου 3 εκατομμύρια επιβάτες χρησιμοποίησαν το εν λόγω τρένο, γεγονός το οποίο μείωσε το χρόνο ταξιδίου μεταξύ Γκάρδης και Παρισίων ε, στις 3 ώρες και 45 λεπτά. Αυτό είναι ήδη κάτω του μαγικού ορίου των τεσσάρων ωρών που είναι το όριο στο οποίο οι άνθρωποι κάνουν την επιλογή μεταξύ τρένου και αεροπλάνου και φαίνεται ότι αυτή η σιδηροδρομική γραμμή ουσιαστικά αντικατέστησε όλες τις πτήσεις μεταξύ Σουτγκάρδης και Παρίσιου και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ένα άλλο καλό νέο είναι το γεγονός ότι το δεύτερο τμήμα του TGV στην Γαλλία μεταξύ Μποντρεγκούρ και Βάντενχάιμ έχει μια επιτυχή οικονομική συμφωνία, υπεγράφει ήδη και θα είναι σε λειτουργία στις αρχές του 2016 η συγκεκριμένη γραμμή. Ένα άλλο κανόν νέο είναι ε, ο νέος κεντρικός σταθμός ε, για τη Βιέννη. Ξεκίνησαν οι εργασίες στις αρχές του έτους και αυτός ο νέος σιδηροδρομικός σταθμός θα μειώσει το χρόνο ταξιδίου κατά 40 λεπτά. Αυτή είναι η μεγαλύτερη χρονική εξοικονόμηση σε όλη την γραμμή και σε όλες τις κατασκευές. Υπάρχουν επίσης κάποιες άλλες σημαντικές ε, ε ημερομηνίες. Υπάρχει μια νέα γέφυρα σιδηροδρόμων στο ποταμό Ρήνο, στο τμήμα ε, Μόναχο Φράιλασινγκ και θα ολοκληρωθεί του χρόνου αυτή η γραμμή. Το Δεκέμβριο φέτος θα ανοίξει η νέα γέφυρα του Κιλ που ήταν ο σύνδεσμος που έλειπε μεταξύ Γερμανίας και Γαλλίας και μία νέα γέφυρα ε, στην οποία μπορεί να υπάρχει ταχύτητα 160 χιλιόμετρων την ώρα. Στη Βαβαρία τώρα, το τμήμα Amfink Mulder θα ανοίξει το Δεκέμβριο φέτος οι εργασίες είναι παραδειγματικές και εν εξελίξη και το τμήμα προς τη Βιέννη φαίνεται ότι θα ολοκληρωθεί μέχρι το 2015. Υπάρχει και ένας νέος σταθμός στο Σάνκ Πούτεν, ο οποίος εγκαινιάστηκε πριν από μερικούς μήνες και το τμήμα Σάνκ Πούτεν Βιέννη θα ολοκληρωθεί μέχρι το Δεκέμβριο του 2012, γεγονός το οποίο θα μας επιτρέψει να μειώθουμε ακόμα περαιτέρω το χρόνο ταξιδίου κατά 15 λεπτά και θα ξεκινήσει και η πολύ σημαντική σύνδεση μεταξύ Βιέννη και Μπρατισλάβα. Αυτό στι αρχέ του νέου έτου. Αυτά είναι τα καλά νέα. Έχουμε βέβαια και κάποιε καθυστερήσει. Το Kiel, Appenweier, Freilancing και η περιοχή των συνόρων έχει καθυστερήσει. Το συναλλικό κόστος ε, του ε, προγράμματος προτεραιότητας 17 είναι περίπου 27 δις ευρώ. Μέχρι το τέλος της προηγούμενης χρονιάς, του 2009, το 50% αυτού του, ποσοστό είχε ήδη, ε, του ποσού είχε ήδη δαπανηθεί. Γεγονός που είναι και πάλι καλό αποτέλεσμα. Θεωρώ ότι με συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε πετύχει πολύ καλή συγκέντρωση, έχουμε καταφέρει να προετοιμάσουμε τα σημεία διάσκησης των συνόρων. Σας ανέφερα ήδη τις δύο γέφυρες, τη μία μεταξύ Αυστρίας και Γερμανίας και την άλλη μεταξύ Γερμανίας και Γαλλίας. Και ε, υπάρχουν και ε, βοήθεια για να μπορέσουμε να ε, επιλύσουμε και κάποιες χερσαίες ε, προβληματικές περιοχές. Επίσης έχουμε χρηματοδότησει μελέτε μέχρι το 15%. Ε, στο παρελθόν είχαμε συμμετοχή στις μελέτες από 44% έως 50% και έχουμε και επενδύσει μεταξύ 3% και 25%. Που και πάλι είναι πολύ σημαντική συνεισφορά. αν προσπαθήσουμε τώρα να κάνουμε μία πρόγνωση, η προθεσμία για τις δημοσιονομικές μας προοπτικές είναι το 2014. Η καταληκτική προθεσμία είναι αυτή και κάναμε έναν υπολογισμό για το τι ακριβώς μας απομένει πέραν του 2014. Ε, από τους υπολογισμούς μας μας απομένει το 21% των επενδύσεων και το 6% των εργασιών. Επομένως, ε, μικρότερο μερίδιο εργασιών και περισσότερα χρήματα τα οποία θα πρέπει να καταβληθούν μετά από το 2014. Πρόθεσή μου είναι να ανανεώσουμε την ε, προθυμία και την ενότητα των κρατών μελών και αυτό το χρειαζόμαστε για δύο βασικούς λόγους. Καταρχάς, ε, διότι οι οικονομικές συνθήκες αλλάζουν βαθμιδών και ε, ε, σε κάποιες περιπτώσεις επιδεινώνονται και επομένως στις νέες προοπτικές θα μπορούσε να γίνει επαναξιολόγηση των προγραμμάτων σε κάποιες χώρες μέλη οι οποίες θα λάβουν υπόψη τις νέες συνθήκες και φυσικά υπάρχει και η αλλαγή των κυβερνήσεων το οποίο είναι φυσική συνέπεια του δημοκρατικού βίου αλλά ε, από τότε που ασχολούμαι εγώ με το πρόγραμμα αυτό ε, με μία μικρή διακοπή έχουμε ένα διάστημα πέντε ετών κατά μέσο όρο τρεις υπουργοί έχουν αλλάξει σε κάθε κράτος μέλος, οπότε χρειάστηκε να ξαναλλάξουν οι εργασίες με κάθε νέα κυβέρνηση, νέο υπουργό, το οποίο είναι φυσικό μεν, προσπαθώ πάντα να το εντάξω αυτό. Ε, βρίσκομαι σε μια δύσκολη θέση μεταξύ των συντονισμών. Ε, με μία διακοπή ε, ήμουνα στην εθνική κυβέρνηση, μετά ξαναδιορίστηκα. Δεν, μπόρεσα να, να, δεν μπορώ να ρίξω το φταίξιμο στον προκάτοχό μου, γιατί εγώ ήμουν ο προκάτοχός μου και αν ε, ε, αποτίσω φόρο τιμή στον προκάτοχό μου θα είναι σαν να ευλογώ τα γένια μου. Ευχαριστώ πολύ. Στη συνέχεια, ο κύριος Μπρίνκχαρς, ο οποίος είναι από το πρόγραμμα προτεραιότητας 6. Ένα πρόγραμμα που αφού ενδιαφέρει το Κοινοβούλιο. Κύριε Πρόεδρε, ελπίζω να μην ε, γίνουμε δίκτυο των πρώην. Δεν ήταν αυτός ο στόχος. Ε, κύριε Πρόεδρε, δεν θα επαναλάβω όλα όσα είπαν οι συνάδελφοι, αλλά... Προφανώς ε, όσον αφορά το πρόγραμμα 6 βρισκόμαστε και εδώ σε κρίσιμη φάση. Δεν χρειάζεται να σας πω ότι είναι η βασική γραμμή Ανατολής Δύσης. Και πολιτικά νομίζω ότι είναι σημαντική διότι έχουν εκφραστεί αμφιβολίες στο Κοινοβούλιο όσον αφορά την πραγματοποίηση. Ε, αλλά η πολιτική δέσμευση δηλώθηκε ρητά όταν συναντηθήκαμε πέρσι στην Σαραγώσα. Οι εμπλεκόμενες χώρες μαζί με τον Επίτροπο έχουν ε, υπογράψει άλλη μία σύμβαση για να προχωρήσουν διότι ε, είναι σημαντικό στοιχείο όχι μόνο για τις χώρες αυτές αλλά και για την Ισπανία και την Πορτογαλία στα δυτικά και ε, για χώρες όπως η Ουκρανία στα ανατολικά. Είναι λοιπόν στρατηγικό σύνδεσμος. Από πολιτικής πλευράς λοιπόν ε, πιστεύω ότι μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει η δέσμευση ε, όπως γνωρίζετε όμως και όπως είπαν οι συνάδελφοι ε, ε, και ως πρώην υπουργό ε, Υγείας ε, πρέπει να πω ότι μου άρεσε η παρομοίωση που έκανε ο Πάτρικ Κόξ για το αυγό και την κότα και τον μπέικον. Όλα συνδέονται μεταξύ τους. Το βασικό θέμα όμως είναι η μη τήρηση των προθεσμιών. Η πρόοδος ήταν άνηση. Θα ήθελα να επικεντρωθώ σε δύο σημεία κλειδιά, διότι έχουμε την περίπτωση Λιών Τωρίνου και μετά από το τούνελ της Γκόθα με 55 χιλιόμετρα ε, θα είναι ε, το δεύτερο μεγαλύτερο τέτοιο έργο και είναι ε, φυσικό να υπάρχουν προβλήματα. Και έχουμε και από την άλλη πλευρά την Τεριέστη. Ήτανε άνηση η πρόοδο, διότι από τη γαλλική πλευρά έχουν ε, πάει πολύ καλά τα πράγματα. Υπάρχουν τρία διερευνητικά τούνελ. Θα βρείτε τι λεπτομέρειε ε, στην έκθεση. Έχουν, όλα, θα, έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλο τη χρονιά αυτή. Και επίση ε, σημαντικό για, τα, για είναι ότι έχει βελτιωθεί η ιστορική γραμμή. Μεγάλο μέρο των επικρίσεων του ε, Κοινοβουλίου ήταν ότι δεν θα το χρειαστούμε διότι δεν είναι αποδοτική η ιστορική γραμμή. Ε, πριν από πάνω από 3,5 χρόνια ξεκίνησα ε, με τη δουλειά αυτή, ταξίδεψα μέσα από τη διαδρομή αυτή ε, και γνωρίζω τις δυσκολίες. Έχει διαβρυνθεί λοιπόν το τούνελ και μέχρι το τέλος χρονιάς θα έχουμε πρόοδο. Από την ιταλική πλευρά είναι διαφορετικά τα πράγματα. Είναι σαφές όμως ότι η Ιταλική κυβέρνηση έχει επιβεβαιώσει και νομίζω ότι αυτό από μόνο του είναι στοιχείο κλειδί. Έχει επιβεβαιώσει λοιπόν η Ιταλική πλευρά ότι μέχρι το τέλος της ε, χρονιάς αυτής ε, θα υπάρχει το τούνελ Μαντελένα, το πρώτο διαρευνητικό τούνελ ε, από Ιταλικής πλευράς. Βρισκόμαστε σε κρίσιμη φάση διότι στο τέλος της χρονιάς η συνθήκη του Τωρίνου του 2001 θα πρέπει να ανανεωθεί ώστε να περάσουμε από την προπαρασκευαστική φάση στην εφαρμοστική. Και όσον αφορά τη χρηματοδότηση, έχει δημιουργηθεί ένα θέμα ανάμεσα στην ε, γαλλική και την ιταλική κυβέρνηση. Και εδώ γίνεται συζήτηση. για το θέμα του κατά πόσο η χρηματοδότηση θα παρατεθεί από την Ιταλική πλευρά. Και φυσικά η κατάσταση του προϋπολογισμού στα κράτη-μέλη, θα συμφωνήσετε όλοι, είναι θέμα ανησυχητικό. Με βάση λοιπόν αυτά, το τέλος της χρονιάς αυτής θα αποτελέσει ε, χρονικό σημείο κλειδί. έχει ζητηθεί για το διάστημα 2013-2014 από ε, τα κράτη-μέλη Ιταλία και Γαλλία να συμφωνήσουν για την ε, χρηματοδότηση. Δεύτερον, ε, να οριστεί νέος προωθητής και να υπάρχει και νέα δομή διαχείρισης για τον φορέα αυτών. Ε, έχει συμφωνηθεί για πρώτη φορά ότι η Κομισιόν θα είναι πλήρης εταίρος, δεν θα είναι παρατηρητής, ε, θα είμαστε εταίρος στην ε, δομή διακυβέρνησης και νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό στοιχείο. Όσον αφορά το άλλο διασυνοριακό τμήμα, πρόσφατα ήμασταν στην Σλοβενία, έχει υπογραφεί συμφωνία ανάμεσα στην Ιταλία και τη Σλοβενία ε, για το ε, κομμάτι τεριέστη τριβάτσα. Αυτό σημαίνει ότι από τη μία θα υπάρχει ε, κοινός Ιταλοσλοβανικός φορέας στην Τεριέστη που θα είναι προκάτοχος της Ευρωπαϊκής Ομάδας Ενδιαφέροντος που θα δημιουργηθεί ε, της οποίας ε, θα είναι ε, και η Κομισιόν πλήρες μέλος. Σημειώστε ότι η Κομισιόν θα είναι και πάλι πλήρως, πλήρες μέλος. Μέρος του διασυνοριακού αυτού κομματιού θα χρηματοδοτηθεί με τα διαρθρωτικά ταμεία. Η διαδρομή αυτή συνεχίζεται μέχρι τη Λιουμπλιάνα και η ε, πρόοδος στο σημείο αυτό είναι επίση ικανοποιητική. Η Σλοβενία ε, έχει δηλώσει ότι το έργο μπορεί να ολοκληρωθεί μέχρι το 2017. Ένα πρόβλημα το οποίο συνδέεται και με αυτό που είπε ο συνάδελφος του Ολιβιέρα ε, είναι ο σύνδεσμος με τα λιμάνια. Η Βόρεια Αδριατική έχει πολύ καλά λιμάνια και θα πρέπει να συνδεθούν και αυτά με το δίκτυο στο κάτω-κάτω. Η συνεργασία ανάμεσα στα, στους δύο αυτούς ε, λιμένες είναι στοιχείο κλειδί για την ε, Βόρεια Αδριατική. Πολύ σύντομα, κύριε Πρόεδρε, όσον αφορά τα δύο εθνικά κομμάτια. Το κομμάτι εντός της Ιταλίας προοδεύει καλά. Πριν δύο εβδομάδες βρέθηκα στην Τεριέστη και ο πρόεδρος ε, ε, της ε, Βένετο και της Γιούλια είχαν συμφωνήσει όσον αφορά την ευθυγράμμιση. Οι δυσκολίες λοιπόν θα ξεπεραστούν και πιστεύω ότι αυτό είναι πολύ θετικό βήμα πρόοδου. Τέλος κύριε πρόεδρε να συνοψίσω. Πρώτον, έχει φτάσει η ώρα της αλήθειας. Στο τέλος της χρονιάς θα πρέπει να ανανεωθεί η συνθήκη της, του Τωρίνου. δεύτερον, όσον αφορά Ε, το, το σύνδεσμο από την ε, Τεριέστη έχει σημειωθεί πρόοδο στη σλοβενική πλευρά και τέλος δεν με ακούσατε να μιλάω για την Ουγγαρία ε, και τα εθνικά κομμάτια εντός της Ουγγαρίας επίσης προχωρούν γρήγορα αλλά το Το Νοέμβριο θα πάμε στην Ουγγαρία για να δούμε κατά πόσο αυτά θα, τα κομμάτια θα συνδεθούν με τα κομμάτια εκτός της Ουγγαρίας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ρίγκορστο. Ο έσκατος Ελλάσσον, ο κύριος Βίνκ. Κύριε Πρόεδρε, μέλη του Κοινοβουλίου, για να συνεχίσω την ε, παρομοίωση που έκανε ο Πατ Κόξ με την κότα και το αυγό θα έλεγα και εγώ ότι συμφωνώ. Το θέμα αυτό έχει συζητηθεί εκτενώς, αλλά υπάρχουν και ορισμένα υποθέματα που θα ήθελα να θίξω. 3.300 χιλιόμετρα ε, ε, ε, χρησιμοποιούνται με το TMS στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να πω ότι έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδο σε ό,τι αφορά τον εξοπλισμό, το DMS που δίνεται από διάφορους προμηθευτές στην Ισπανία, την Ιταλία, την Ελβετία και την Ολλανδία. Αν διαβάσατε την ενδιάμεση έκθεση θα έχετε διαπιστώσει ότι υπάρχει μια πάρα πολύ, καθίστε απόλυτα σαφής η πολιτική αυτή και θα είναι ακόμα σαφέστερη στο μέλλον πιστεύω. Κάτι που θα ήθελα να τονίσω και να υπογραμμίσω είναι ότι αυτό γίνεται το σήμα κατά τεθέν έξω από την Ευρώπη. Υπάρχουν πάνω από 10.000 ε, χιλιόμετρα που έχουν εξοπλιστεί με TMS εκτός Ευρώπης, Σαουδική Αραβία, ε, Κίνα ε, και πραγματικά είναι ένας πολύ μεγάλος παράγοντας τον ηγετικό ρόλο που παίζουμε στην Ευρώπη και θα πρέπει να τον υποστηρίξουμε γιατί είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα από την τεχνολογία. Ε, Εάν θέλουμε όμως να προχωρήσουμε θα πρέπει να ασχοληθούμε με μία σειρά από θέματα. Το ένα είναι η εναρμόνιση και η απλοποίηση του δικτύου. Το δεύτερο είναι τα προβλήματα που έχουμε για την ώρα στη Γερμανία. Η Γερμανία είναι πολύ σημαντική γιατί βρίσκεται στο μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το τρίτον, η μείωση που απαιτείται σε επίπεδο κόστους, μιλώντα για εξοπλισμό ε, ε, ε, RTMS. Δύο λόγια για την εναρμόνιση και την απλοποίηση του RTMS. Από τον Ιούλιο του 2008 και την υπογραφή της συμφωνίας έγιναν πολλές, στη Ρώμη έγιναν πολλές συζητήσεις και πολλές συνεργασίες μεταξύ της Επιτροπής, της ΕΡΑ και των βασικών ε, συντελεστών. Πρόσφατα εξετάσαμε τη δυνατότητα να επιταχύνουμε τον ρυθμό ανάπτυξης του ε, ε, ERTMS. Ε, υπάρχει λοιπόν μια σειρά από συστάσεις και τα όσα θα σας πω τώρα αναφέρονται στα συμπεράσματα ε, αυτών των συστάσεων. Καταρχάς εναρμόνιση. Θα ήθελα πρώτον να τονίσω τα λειτουργικά θέματα. Όταν ξεκινήσαμε είπαμε ότι χρειαζόμαστε τρία πράγματα για να μπορέσει να λειτουργήσει αυτό το σύστημα διαχείρισης των χερσαίων μεταφορών, το, το RTMS. Να βελτιώσουμε τις υποδομές, να εισαγάγουμε το RTMS και να ε, βελτιώσουμε τους κανόνες. Καταλαβαίνουμε, λόγω των περιορισμών του προπολογισμού και σε επίπεδο χωρών μελών, αλλά και σε επίπεδο επιτροπής, ότι θα μπορούσαμε να τα αντιστρέψουμε τα πράγματα. Δηλαδή θα μπορούσαμε να κοιτάξουμε τον, ε, την εναρμόνιση των κανόνων γιατί αυτό είναι ένα θέμα βούληση μεταξύ των χωρών μελών και τη επιτροπή και δεν κοστίζει και τόσα πολλά χρήματα. Το θέμα είναι πόση επιθυμία έχουν, πόση βούληση υπάρχει. Βεβαίω υπάρχουν ορισμένα πράγματα που εύκολα θα μπορούσαν να γίνουν. Καταρχά το μήκος των τρένων. Κατά μέσον όρων είναι 440 μέτρα. Δίχω σημαντικές επενδύσεις θα μπορούσαμε να φτεράσουμε στα 750 μέτρα. Αυτή είναι μια άμεση αύξηση της παραγωγικότητας. Αυτή είναι μια καλύτερη λύση στο πρόβλημα των μεταφορών. Από αυτή την άποψη λοιπόν, θα έλεγα γιατί δεν το κάνουμε. Υπάρχουν και άλλα πράγματα που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Το βάρο η λειτουργική ταχύτητα, η, η πολλά μέτρα που δεν κοστίζουν κοστίζουν πάρα πολλά αλλά που συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα των ε, μεταφορών. Ένα άλλο θέμα που θα ήθελα να τονίσω την εναρμόνιση των διαδικασιών ε, έγκρισης. Οι διαδικασίες έγκρισης αποτελούν ένα σημαντικό πρόσκομα στη διαδικασία αυτή. Στην ουσία υπάρχει ένας φαύλος κύκλος που θα πρέπει να σπάσει ε, τα προαπαιτούμενα αλλάζουν από τη μία χώρα στην άλλη. Και μετά βεβαίως υπάρχουν αδυναμίες στον εξοπλισμό. Συνεπώς η διαδικασία των αδειών, αδειοδότηση θα μπορούσε να εναρμονιστεί και αυτό θα αποβεί υπέρ του συστήματος μεταφορών. Δεύτερο θέμα η τυποποίηση πέρα από την εναρμόνιση. Πιστεύω ότι πολλές φορές γίνονται πάρα πολλές συζητήσεις σε ό,τι αφορά τις, ε, την τυποποίηση που χρειάζεται. Θα μπορούσαμε να κάνουμε πολλά σε αυτό το τομέα και θα μπορούσα να γίνουμε βάση τα όσα αποφασίστηκαν σε επίπεδο επιτροπής. Έχουμε τώρα τα προτυπα 2 0 3.0D και γίνονται προσπάθειες έτσι ώστε να μπορέσουν να αναπτυχθούν καλύτερα τα ATMS. Ε, Επίσης, το 2012 προβλέπεται ένα άλλο πρότυπο το οποίο το 300 και αυτό θα μπορούσε να ε, εισαχθεί στα έγγραφα των διαγωνισμών. Δεν ε, τυποποιούμε αλλά υπάρχει κατά την άποψή μου μια δυνατότητα που δεν νομίζω να παρουσιάζει προβλήματα. Θα πρέπει να βελτιώσουμε το διάλογο μεταξύ των διαφόρων συντελεστών τις, ε, τους υπεύθυνους ε, για τις υποδομές, ε, τις εθνικές αρχές ασφαλείας που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, αλλά και την, τον Ευρωπαϊκό Εθνικό Φορέα Αν βελτιώσουμε τα πράγματα εκεί, δίχως άλλο θα προχωρήσουμε να προχωρήσουμε. Βεβαίω, και η τυποποίηση. Αυτό είναι ένα πολύ βασικό θέμα. Ένα θέμα που μας απασχολεί ιδιαίτερα και συνεργαζόμαστε με τους ε, κατασκευαστές και που δίχως άλλο θα συμβάλλει στην ανάπτυξη του RTMS. Ε, θα ήθελα επίση να υπογραμμίσω το πόσο σημαντικό είναι να εναρμονίσουμε και να τυποποιήσουμε τη διαδικασία. Σήμερα περνάμε τις διάφορες δοκιμές που προβλέπονται σε διάφορα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρξει μια κοινή διαδικασία δοκιμών. Αυτό είναι ένα σημαντικό μέλος της εντολής μου ως συντονιστή με ενδιαφέρει ιδιαίτερα να υπάρξουν κοινέ διαδικασίες ε, εργαστηριακές θα μπορούσαν να, να εισαχθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο και πιστεύω ότι αυτό θα συνέβαλε πάρα πολύ. Ύστερα έχουμε τον συντονισμό της, ε, των ε, διαφορών επενδύσεων. Τόσα λέμε θα μπορούσαν να συμβούν αν υπάρχει μια συμφωνία μεταξύ των διαφόρων συντελεστών των διαδρόμων έτσι ώστε να γίνει από κοινού και να γίνει και προγραμματισμένα θετικό είναι ότι ιδιαίτερα για του διαδρόμου των εμπορευμάτων υπάρχει μια οργάνωση. Στο ανώτατο επίπεδο έχουμε του υπουργού μεταφορών και τις χώρες μέλη που ε, ε, ε, έχουν σχέση. Μετά έχουμε τον ανώτατο εκπρόσωπο όλων των υπουργών και την Εκτελεστική Επιτροπή η οποία είναι υπεύθυνη για το πρόγραμμα για τον διάδρομο. Σε επίπεδο διαχείριση έχουμε τους υπεύθυνους διαχειριστέ, που είναι υπεύθυνε όχι μόνο για την ανάπτυξη ενό προγράμματο, αλλά και για την εφαρμογή και πραγματοποίησή του. Αυτή η δομή υφίσταται εδώ και τρία χρόνια στο διάδρομο Ρότερνταμ Τζένοβα, στο διάδρομο C και τώρα χρησιμοποιείται και στο βασικό διάδρομο εμπορευμάτων. Έχουμε προδεύσει, έχουμε προδεύσει λόγω αυτής της οργάνωσης και φαντάζομαι ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε και στο μέλλον. Απαιτείται ένα συντονισμός μεταξύ των διαφόρων συστημάτων γιατί δεν μπορούμε να περάσουμε από τη μία στιγμή στην άλλη στο σύστημα RTMS. Απαιτείται λοιπόν ο συντονισμό για να μπορέσουν αυτά να εφαρμοστούν με ένα βέλτιστο τρόπο. Εν συντομία θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο για τη Γερμανία. Η Γερμανία διαδραματίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο. Υπάρχουν τέσσερις διάδρομοι εμπορευμάτων προς τη Γερμανία και υπάρχουν και υπήρχε και μία δέσμευση από πλευράς γερμανικής κυβέρνησης να ληφθούν υπόψη οι εξοπλισμοί που απαιτούνται για τους ε, τέσσερις διαδρόμους. Ε, υπάρχουν παράγοντες που γνωρίζετε και εσείς, όπως και εγώ και το λόγο αυτό, υπάρχουν ορισμένες επιφυλάξεις. Η Γερμανία τράβηξε λίγο το φρένο σε επίπεδο εφαρμογής. Υπάρχει εδώ ο Υπουργό Μεταφορών είπε εντάξει ας ε, καθορίσουμε ως βασική προτεραιότητα το διάδρομο A. έχουμε προχωρήσει αρκετά σε ό,τι αφορά το RTMS. Σε ό,τι αφορά τους άλλους διαδρόμους, ας δούμε τι είναι δυνατόν, λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς όπως παρουσιάστηκαν στη Γερμανία. Και όταν συζητήσαμε με τη γερμανική κυβέρνηση μπορέσαμε να εντοπίσουμε τρεις λόγους για τους οποίους γίνεται αυτή η συζήτηση. Η πρώτη συζήτηση αφορά το κόστος. Θα πρέπει να είμαι απόλυτα σαφής. Υπάρχουν ορισμένες ιδέες που αφορούν το κόστος για την Γερμανία. Ε, ε, ε, έγινε αναφορά σε συγκεκριμένα ποσά σε 4,5 δις. Αυτό βεβαίως για το σύνολο των διαδρόμων. Αν όμως λάβουμε υπόψη τις προτεραιότητες και ιδιαίτερα το διάδρομο Α, τότε τα ποσά είναι πολύ χαμηλότερα και που είναι γύρω στα 450 εκατομμύρια ευρώ σε ένα διάστημα 5 ετών. Κατά την άποψή μου για μια χώρα, για την, ε, σαν τη Γερμανία, αυτό θα μπορούσε να είναι εφικτό και θα μπορούσε να μας ε, ε, δώσει πολλές δυνατότητες, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό σε ό,τι αφορά την διαλειτουργικότητα. Συζήτηση για το κόστος. Θα πρέπει να είμαστε απόλυτα σαφείς σε ό,τι αφορά αυτό το θέμα η συζήτηση για τις τεχνικές λύσεις. Φαντάζομαι ότι γίνονται συζητήσεις για τα διάφορα πρότυπα, αλλά αυτό θα μπορούσε να επιληθεί. Είναι ένα θέμα όμως αρκετά τεχνικό. Μετά η συζήτηση για τη διαθεσιμότητα του προπολογισμού, για τις τεχνικές λύσεις. Δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν αυτά γιατί υπάρχουν περιορισμοί του προπολογισμού όπως επιβάλλονται από τους Υπουργού Οικονομικών λαμβάνοντας υπόψη τα όσα είπα σχετικά με το κόστος σκέφτομαι ότι υπάρχει ένας τρόπος που μας δίνει τη δυνατότητα να συνεχίσουμε με το διάδρομο Α ως πρώτη προτεραιότητα και μετά θα υπάρξει ένα εκτενέστερο χρονικό διάστημα για τους άλλους διαδρόμους εμπορευμάτων. Και το τρίτο στοιχείο, μείωση του εξοπλισμού Αυτό δεν είναι εξοπλισμό του ATM. Ε, θα πρέπει να μας απασχολήσουν και ορισμένα θέματα που αφορούν τις αρκές ασφαλείας. Και εκεί μπορούν να γίνουν απλοποιήσεις και εκεί μπορούν, ε, μπορεί να υπάρξει μία μείωση του κόστους και αυτό με ένα συντονισμένο τρόπο. Το άλλο είναι τι είδους ερέτηση, τι είδους κίνητρο χρειαζόμαστε για να κάνουμε αυτό το πέρασμα. Πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να στοχεύσουμε σε μία έκπτωση 5%. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας, με ένα κόστος επένδυσης 200.000 ευρώ, θα μπορέσουμε να τα καταφέρουμε σε 5 ή 6 χρόνια. Βλέπετε λοιπόν ότι προχωράμε. Είμαι αισιόδοξο σε ό,τι αφορά τις δυνατότητες. Έχουμε μια τεχνική λύση από αυτή την ε, ε, νόμιμη το τεχνικό Υπάρχει ένα, οικονομικό, ένα τεχνικό πρόβλημα, υπάρχει ένα οικονομικό πρόβλημα, αλλά το δυνητικό αυτή της μεθόδου για να επιτευχθεί η βελτιστοποίηση βρίσκεται στα χέρια μας. Βεβαίως υπάρχουν καθυστερήσεις, αλλά είναι υποέλεγχο. Συνεπώς από αυτή την άποψη πιστεύω ότι το μόνο που θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι να συνεχίσουμε ε, και να προχωρήσουμε όπως είπε ο Πάτκο. Ωραία, ευχαριστώ. Τον κύριο Βίνκ και φυσικά τους κυρίους ε, Κόξ, Πάλακ και Brinkhorst. Θα διαβάσω όλου όσου έχω στον κατάλογο. Αν δεν είστε στον κατάλογο και θέλετε να μιλήσετε, να μερώστε με. Sender, Mrs. Lichtenberger, Mr. Urias, Mrs. Fayon, Mr. Kuhn, Mr. Rike, and Mr. Bach. Mr. Cock, I've seen anybody else. Δεν βλέπω κάποιον άλλον, επομένως ε, θα προχωρήσουμε έτσι. Ο κύριος Καντσιάνη καταρχάς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι που σήμερα άκουσα τους τέσσερις συντονιστές οι οποίοι παρουσίασαν ε, κάποια πάρα πολύ σημαντικά θέματα για το ΕΛΚ. Νομίζω ότι η ναυαρχίδα, κύριε Κόξ, είναι το σύνολο αυτών που ακούσαμε σήμερα εδώ έχουμε δύο διαδρόμους, τον 17 και τον 6, ο ένας από τη μια και ο άλλος από την άλλη πλευρά των Άλπαιων, που συνδύονται με το πρόγραμμα προτεραιότητας 1, καθέτος και αν δούμε προς δυσμάς, το Γένοβα, Ρότερνταμ και προς Ανατολάς ε, πάμε από τον P6 ε, μέχρι επάνω, ουσιαστικά έχουμε ένα ουσιαστικό δίκτυο, σημαντικό δίκτυο ανάπτυξης Ευρώπης μας. Θεωρώ λοιπόν ότι σήμερα βρισκόμαστε στο επίκεντρο των θεμάτων που αφορούν τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Αυτό, από, κατά την άποψή μου, μαζί με τη σωστή χρήση και τη σωστή διαχείριση του RTMS, δηλαδή αυτό του συστήματος διαχείρισης, το οποίο με τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη για να ξέρουμε ποιο είναι αρμόδιος γιατί. Θεωρώ ότι πρόκειται για το τέλειο πλαίσιο και φρονώ επίση ότι από πολιτική πλευρά δεν θα πρέπει να οπισθοδρομούμε, αλλά θα πρέπει να βλέπουμε προ το μέλλον. Αυτό είναι το όρομα που έχουμε εμεί σήμερα και θεωρώ ότι θα πρέπει να εκτιμήσουμε τα όσα έχουν γίνει μέχρι τούδε, διότι εγώ Είχα και τη δυνατότητα να μιλήσω και με τον κύριο Κόξ και με τον κύριο Μπρίνχοστ ε, σε συγκεκριμένες ε, περιπτώσεις και ξέρω ότι ε, δεσμεύτηκαν προκειμένου να προχωρήσουν αυτές οι εργασίες από τις ε, εκθέσεις τους. Διαβάζω μεν για κάποιες καθυστερήσεις, για κάποια προβλήματα, αλλά ε, διαπιστώνω ότι υπάρχει και μία αισιοδοξία και θα ήθελα να επαναλάβω εδώ ότι δεν θα πρέπει να χάσουμε ποτέ την αισιοδοξία μας. Διότι μπορεί να υπάρξουν κάποια σημεία που μπορεί να υπάρχουν προσκόμματα ε, σε ένα τέτοιο πρόγραμμα και εάν σταματήσει αυτό δεν κάνουμε κακό μόνο στη συγκεκριμένη περιοχή αλλά κάνουμε συλλογικό κακό σε ένα ε, ευρωπαϊκό σχέδιο αυτή είναι η άποψή μου και νομίζω και όλου του ΕΛΚ, γιατί μιλώ και εξ ονόματος του ΕΛΚ. Αυτό το οποίο θα ήθελα να επαναλάβω είναι το εξή. Εάν ε, διαβάσουμε το βαθύτερο νόημα της έκθεσης που μας έκανε ο Επίτροπος, ε, η έλλειψη χρηματοδότηση ε, πηγαίνει αρνητικά στα ήδη υφιστάμενα προβλήματα και δεν είναι αυτό ο τρόπος επίλυσης, διότι αν υπάρχουν καθυστερήσει, ορισμένες φορές υπάρχουν γραφειοκρατικά προβλήματα, τοπικά προβλήματα, αλλά το βασικό πρόβλημα είναι η έλλειψη συγχρηματοδότηση. ιδίω τώρα που έχουμε κρίση. Αυτό είναι ο πραγματικό ε, γόρδιος δεσμό που έχουμε να λύσουμε αυτή τη στιγμή. Δεν πρέπει λοιπόν να σταματήσουμε την χρηματοδότηση, αλλά πρέπει να συνδράμουμε για να επιληθεί το πρόβλημα. Επίσης, πρέπει να δούμε και τι εξουσία έχουν οι συντονιστές αυτοί να μπορέσουν να προχωρήσουν τα θέματα και να προσπαθήσουν να λύσουν κάποια τοπικά προβλήματα, διότι αν βρεθεί κάποιο επιτόπου ε, μπορεί να έχει πρόβλημα. Αλλά ο Επίτροπος ο οποίος βλέπει το θέμα ευρωπαϊκά μπορεί να μπορέσει να λύσει και πιο εύκολα. Δεν ξέρω ακριβώ πώ, αλλά να το έχουμε κατά νου και αυτό για να μπορέσουμε ίσως να διευκολύνουμε αυτή την κρίσιμη περίοδο που μπορεί να ζήσει κάποιο επιτόπου σε, μια περιοχή. Θεωρώ ότι αυτή είναι η σωστή άγουσα. Αυτός είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε. Και θεωρώ ότι ο Επίτροπος ο οποίος ε, αφενός μας παρουσίασε τι προβλήματα σχετίζονται με τη χρηματοδότηση Νομίζω ότι υπάρχει δυνατότητα να παρέμβουμε ε, όχι μόνο μέσω προπολογισμού, αλλά δίνονται και άλλες δυνατότητες να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι ώστε πέραν των μελετών σε κάποιες περιπτώσεις να υπάρχει δυνατότητα να υλοποιήσουμε και κάποια πράγματα. 8 δις ε, αντί 500 ε, που μας υπόθηκε νομίζω ότι σημαίνει ότι πρέπει να βρούμε και έναν τρόπο να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα για το μέλλον. Η κυρία Γιάλα Σέντερ για τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να θέσω από μία ερώτηση σε κάθε ένα από τους συντονιστές. Τους ευχαριστώ, όπως έλεγε και ο συνάδελφος, ε, για το αισιόδοξο πεδίο που μας παρουσίασαν ε, και το παράδειγμα με το γουρούνι και την κότα. Εγώ δεν ξέρω ποιος είναι ποιος, αλλά τέλος πάντων το παράδειγμα μας έδωσε και κάποια εικόνα. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξή. Η μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση, η ερώτηση είναι και προ του τέσσερι ή τουλάχιστον προ του τρει που ασχολούνται με σιδηροδρόμου, με συγκεκριμένου διαδρόμου. Στα προγράμματά σα εκκρεμούν ε, αυτές οι προϋποθέσεις που τίθενται από το η μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση, αυτό το έγγραφο που μόλις λάβαμε, υποθέτω ότι λάβατε κι εσείς, σας βοηθά ή δεν σας βοηθά στην επικοινωνία με τις διάφορες περιοχές και τους υπεύθυνους και τους ε, χορηγούς. Διότι στο πρόγραμμα 1 αναφέρεται σαφώς ότι το νότιο τμήμα θα έχει προβλήματα, ε, το τμήμα του Μπρένερου θα έχει προβλήματα. Στον κύριο Μπάλας και ήθελα να ρωτήσω το ίδιο πράγμα. Θεωρείτε και εσείς ότι η τεχνική λύση για τη στροφή της Καρλουέ ε, θα έχει αποφασιστεί πριν από το τέλος του 2010, διότι είναι το πρόβλημα το οποίο προκύπτει για να συνεχίσει η χρηματοδότηση τμήμα του προγράμμα, ε, τμήματος του προγράμματος που έχετε εσείς. Τώρα, για το Λιόν ε, το Ρίνο που το παρακολουθώ λες και είναι αδελφός σιδηρόδρομος του Ισπανικού προγράμματος, θεωρώ ότι οι Ισπανοί και οι Πορτογάλοι θα υποβαληθούν διότι θα μπορεί κάποιο να φτάσει και από Ισπανία ε, στη Λιόν για να πάρει και το σιδηρόδρομο Λιόν Τουρίν ε, και για την κεντρική γραμμή των PP16. Ε, θα ήθελα να ρωτήσω το ίδιο. Οι νέε προϋποθέσεις που προκύπτουν από την μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση σας βοηθούν? Διότι ειδικά στο πώ ε, θα καθοριστεί ο σχεδιασμός κάποιων προβλημάτων ε, στο διεθνέ κομμάτι είναι πολύ σημαντικό, Κυρίω για το Λιόν το πριν από το 2016. Κύριε Μπριγχόρστ, όπω γνωρίζετε, η Ισπανία θεωρεί ότι η σιδηρόδρομοι αυτή είναι μία από τους άξονε ένας από τους άξονες προτεραιότητας. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι που είναι ενδιαφέρον για κάθε αναδιατύπωση των σιδηροδρομικών πακέτων. Η εφαρμογή του RTMS θα έχει και μείωση στο κόστος για τις σιδηροδρομικές γραμμές. Ευχαριστώ κυρία Μάισνερ και τους φιλελευθέρους. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά και εγώ τους συντονιστές. Είναι πολύ σημαντική η σημερινή ημέρα διότι μαθαίνουμε πολλές λεπτομέρειες σχετικά με τα μεμονωμένα προγράμματα τα οποία κρεμούν. Έτσι μπορούμε να τα κρίνουμε καλύτερα και να οργανώσουμε τη δουλειά μας καλύτερα. Θα ξεκινήσω από τον κύριο Μπρίγχος διότι είναι ο μόνος που δεν αναφέρεται στην Γερμανία. Ε, δεν γνωρίζω πολύ καλά το έργο σας, γι' αυτό η ερώτησή μου είναι ε, υπό το φως ότι είπατε ότι μέχρι το 2015 οι χώρες έχουν χρόνο να δείξουν ότι επικεντρώνονται στο θέμα και ότι συνεργάζονται. Πιστεύετε ότι διακυβεύεται κάτι, εάν ναι, τι και τι μπορούμε να κάνουμε για να ε, διευκολύνουμε το έργο. Διότι από Τη μία θέλουμε να δούμε πώ θα πάνε τα χρήματά μα, από την άλλη θέλουμε να ολοκληρώσουμε το ε, ε, ευρωπαϊκό δίκτυο. Να να ξεκινήσω από τον κύριο Κόξ. Είπατε ότι δεν συμβαίνουν πολύ καλά πράγματα στη Γερμανία. Μπορείτε να μας πείτε τι, ε, τι μπορούμε να ε, κάνουμε για να βοηθήσουμε, διότι ναι, ε, είμαστε Γερμανοί. Θέλουμε όμως να βοηθήσουμε και στην ε, ολοκληρώση και στην ανάπτυξη των διευρωπαϊκών δικτύων. Κύριε Μπάλλας, μια συγκεκριμένη ερώτηση, λίγο καυτή. αναφερθήκατε στον διάδρομο 17 και γνωρίζετε ότι αυτή τη στιγμή στη, το, γνωρίζετε το, το ε, έργο Στουτγάρδη 21 και ξέρετε ότι εκεί έχουν γίνει πολλές διαμαρτυρίες. Πόσο θα διευκολυνθεί το δίκτυο αυτό υψηλής ε, ταχύτητας ε, και πόσο, ε, πόσες εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα μπορούμε να γλιτώσουμε με το σύστημα αυτό. Και πιστεύετε ότι μπορεί να, να τίθεται σε κίνδυνο το έργο λόγω των διαμαρτυριών και να ξεκινήσω και πάλι από τον κύριο Πάλλας για την τελευταία ερώτηση. Είπατε ότι η Γερμανία βρίσκεται στη μέση. Ε, εδώ μπορούν να προχωρήσουν πολλά καλά προγράμματα. Είπατε επίσης ότι η γερμανική κυβέρνηση εν μέρη έχει ε, λάθος παραστάσεις σχετικά με το πόσο θα στοιχήσει. Έχετε συγκεκριμένα έργα τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να συνεχιστεί η σχετική συζήτηση στη Γερμανία. Ευχαριστώ πολύ απελπισμένα προσπαθώ να μην γίνει μια συζήτηση μεταξύ εξήγια. δεν τα κατάφερα. Κύριο Κράμερ. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο παρότι είμαι Γερμανός. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συντονιστές ε, Καταρχήν, κύριε Κόξ, ε, παρουσιάσατε πολύ αισιόδοξα τα πράγματα, ε, αλλά η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Ε, η Νιρεμβέργη Ερφούρτ έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί το 2010. Αν είμαστε τυχεροί, το 2017 θα ολοκληρωθεί, αν όχι το 2020, όσον αφορά το τούνελ του Πρενέρο. Έχουμε δύο τούνελ ήδη το ένα έχει ολοκληρωθεί, το, στο άλλο έχουμε προχωρήσει καλά, αλλά συνεχίζεστε να ε, επικεντρώνεστε στο τούνελ του ε, Πρενέρο, χωρίς να ξέρετε πώς ε, είναι οι δρόμοι προσέγγισης στην Γερμανία. Γιατί δεν λέμε ότι εντάξει να ε, ε, συνεχίσουμε τις εργασίες ε, και στα τρία τούνελ. Ναι, θα πρέπει να αλλάξει αυτό. Αναφέρθηκα στους όρου, στις οδούς προσέγγισης στη Γερμανία. Δεν αναφέρατε καθόλου το, τη γέφυρα της Μεσίνα. Ε, δεν ανήκει και αυτό στο πρόγραμμα αυτό. Μπορείτε παρακαλώ να, να αναφερθείτε σε αυτό. Κύριε Μπάλες, δεν αναφερθήκατε καθόλου στο, στη Στουργάρδη 21. Όλος ο κόσμος μιλάει για αυτό. Σε όλες τις εφημερίδες αναφέρεται αυτό. Ο πληθυσμό της του σε ε, διαμαρτύρεται. Γιατί, διότι έχει ε, εκραγεί το κόστος. Εάν όλα τα χρήματα πάνε στην ε, Στουτγάρδη και δεν θα μείνει τίποτα για άλλα έργα, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Και δόξα τω Θεώ πάντα λέγατε και κάθε φορά ρωτώ και σας ευχαριστώ για τις ειλικρινείς απαντήσεις. Το, ο σταθμός της Στουτγάρδη δεν είναι ευρωπαϊκό έργο. Ε, Ποτέ δεν έχει ε, συμφωνήσει το Κοινοβούλιο για το θέμα αυτό, παρότι η κυρία ε, ε, Μέρκελ και πολλοί άλλοι το υποστηρίζουν αυτό. Παρακαλώ, ξαναπείτε το αυτό. Δεν θέλουν να το ακούσουν αυτό στη Γερμανία, ότι δεν είναι ευρωπαϊκό έργο, αλλά πρέπει να το ακούσουμε. Το 70% των ανθρώπων χρησιμοποιούν το σταθμό της ε, Στουτγάρδης. Αλλά δεν είναι δυνατόν να μην λάβουμε η υπόψη μας ε, και τι μετακινήσης ε, αγαθών. Αυτό το λάβαμε υπόψη μόνο κατά την σύγκριση κέρδους κόστους όφελους. Θα έχουμε λοιπόν δύο ε, διασυνδέσει ε, που δεν θα είναι χρήσιμε όμως ε, για την μετακίνηση αγαθών. 7 δισεκατομμύρια έχουν επενδυθεί και σε μια δεύτερη διαδρομή που επίσης δεν, είναι, δεν μπορεί να λειτουργήσει για τη μετακίνηση των αγαθών. Θα πρέπει να βγάλουμε εμεί τα σωστά συμπεράσματα αυτά. Βλέπετε τι γίνεται στη... στο νέο σταθμό της Βιέννης. Έχει γίνει αποδεκτός. Αυτό μπορεί να το καταλάβει κανεί είναι άλλη υπόθεση. Ε, και ε, θα έχουμε νέο σημείο συμφόρηση στην Στουτκάρδη. Όλο αυτό θα είναι εις βάρος ε, των περιφερειακών μεταφορών. Δεν μπορεί να επενδύσουμε δισεκατομμύρια ώστε να δημιουργήσουμε ένα νέο σημείο συμφόρηση το οποίο θα πρέπει να λύσουμε. Κύριε Πρίγκο, αναφερθήκατε στο, στη σύνδεση Λιών-Τωρίνου. Πιστεύετε ότι θα προχωρήσει αυτό. Ωραία αυτά που μας είπατε, αλλά ε, είναι αλήθεια αυτά. Και κύριε Βίνκ, ε, η ε, Γερμανία μπλοκάρει ε, το έργο, προτιμάει να απεμβολήσει 23 εκατομμύρια Είπατε ότι 4,5 δισεκατομμύρια ε, είναι το ποσό, μπορεί να είναι ακόμα περισσότερο στο μέλλον. Ε, είναι ε, ανταγωνιστικό προτέρημα για τις γερμανικές συνδρομικές γραμμές. Τεχνικά υπάρχουν πολλές ασάφειες εδώ πέρα. Είχαμε 20 διαφορετικά ε, συστήματα στην ε, Ευρώπη, τα αντικαθιστούμε με άλλα 20 όμω τα οποία δεν είναι συμβατά μεταξύ τους. Θα πρέπει να είναι σαφέ αυτό και θα πρέπει να πιέσουμε ε, να αναπτύξουμε περαιτέρω το σύστημα. Για παράδειγμα, ο διάδρομος 1 γιατί δεν επεκτείνεται μέχρι το Ρωστό Κοπενχάγη και Στοκχόλμη. Αυτό θα ήταν πολύ καλό αλλά υπάρχει ε, πριν ε, το λιμάνι του Ροστόκ 10 ε, χιλιόμετρα κενό και το ίδιο πριν το Βερολίνο. Αυτό είναι τρελό. Και τελευταία ερώτηση. Όσον αφορά το Περπινιά, οι Γερμανοί δεν θέλουν ερατεμές, οι οι Ισπανοί το θέλουν. Τι θα γίνει με τα τρένα αυτά. Ε, και τέλος, γιατί δεν ε, εναρμονίζουμε ε, τους όρους κατά την ανάθεση των έργων. περιμένω να ακούσω τις απαντήσεις σας. Ευχαριστώ. Μάικολ, από τότε που άρχισες να μιλάς, μεγάλωσε και ο κατάλογος των ομιλητών μου. Εσύ φταίς νομίζω. Υποθέτω ότι έχεις και κάποιες αμφιβολίες για το Stuttgart 21, ε. Αλήθεια λέω. Next. Στη συνέχεια θα κάνω μία απόπειρα. Αν κάποιο θέλει να πει κάτι για τη Στουτγκάρδη 21, να το πείτε στα γρήγορα για να προχωρήσετε. Το πιάσαμε το μήνυμα για τη Στουτγκάρδη 21. Στη συνέχεια, η κυρία Ράνερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω και πάλι να είμαι σύντομη. Θα... Ήθελα ως Αυστριακή να απευθύνω την ερώτημά μου προς τον κύριο Κόξ ε, και έχει να κάνει με το τούνελ ε, Πρενέρο. Ε, μου προκαλεί εντύπωση μετά από ένα χρόνο στο Κοινοβούλιο γιατί ε, ο καθένας εκπλήσεται με το πόσο ακριβά είναι τα έργα υποδομής. Ε, δεν μπορούμε να τα πληρώσουμε αυτά με έναν πραχυπρόθεσμο προϋπολογισμό. Πρέπει να τα σχεδιάσουμε πιο μακροπρόθεσμα. Ε, και αυτή τη στιγμή στην Αυστρία συζητιέται ο προϋπολογισμός της επόμενης χρονιάς και αυτό δεν αφορά ε, μόνο το τούνελ ε, brenner Μπάζε. Θα ήθελα να σας ευχηθώ ε, κάθε επιτυχία στις διαπραγματεύσεις σας με την Ιταλία. Σας εύχομαι επίσης δημιουργικότητα και αντοχή. Ακούγεται ότι υπάρχουν γεωλογικές δυσκολίες στο τούνελ του Πρενέρο, ε, όπως επίσης και στους ε, δρόμους πρόσβασης. Μπορείτε παρακαλώ να μας πείτε μερικά πράγματα γι' αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Ράνερ. Η κυρία Λίχτεμπέργκερ στη συνέχεια. Φαντάζομαι ότι ξέρω τι ακριβώς θα σας ρωτήσει η κυρία Λίχτεμπέργκερ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ να ζητήσω συγγνώμη. Μπαινοβγαίνω, έχω ταυτόχρονα την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Είναι πολύ δύσκολο αυτό. Ε, δεν άκουσα πλήρως όλες τις, ε, εισηγήσει σα. σας, ε, διάβασα όμως ε, κάποια πράγματα. Αναφέρεται σαφώς ότι, και απευθύνομαι στον κύριο Κόξ καταρχήν, εάν δεν διασφαλίζονται οι βόρειοι και νότιοι δρόμοι πρόσβασης, τότε θα πρέπει να αμφισβητηθούν ε, τα προγράμματα. Κατά τη γνώμη μου, ε, ο νότιος ε, δρόμος πρόσβασης στο τούνελ Πρενέρο δεν πρέπει να αμφισβητηθεί. Το αναφέρετε και εσείς στην έκθεσή σας. Δεν υπάρχει ούτε σχετικό πρόγραμμα και αν ξέρουμε πόσο χρόνο παίρνει στην Ιταλία η υλοποίηση ενός προγράμματος, το πόσο μεγάλο διάστημα μεσολαβεί από το σχέδιο μέχρι το έργο, θα πρέπει να εξετάσουμε την υπόθεση επίσης. Ε, ξέρουμε ότι ένα τούνελ συνδρομικό στην Ιταλία είναι πολύ πιο ακριβό στην Ιταλία από ό,τι στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτό προκύπτει στατιστικά από ε, έργα που ήδη έχουν πραγματοποιηθεί. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να κάνουμε εδώ την διάκριση ανάμεσα σε γεγονότα και υποσχέσεις. Δεν υπάρχουν ούτε σχέδια ακόμα. Οι υποσχέσεις είναι ότι ίσως κάποια στιγμή να βρεθούν χρήματα στην Ιταλία ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τα έργα αυτά. Παρακαλώ λοιπόν να εξετάσουμε και εναλλακτικά έργα προτού να ασκήσουμε πίεση για το θέμα αυτό. Κύριε Μπάλλας. Ε, ένα πολύ ωραίο διάδρομο πέρα από κάποιες μικρές δυσκολίες. Ε, θα ήθελα όμως ε, να επαναλάβω μια ερώτηση που πάντα θέτω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, να δημιουργήσουμε ένα βιομηχανικό τρίγωνο να μην έχουμε έναν ε, άξονα νότια του ε, Σαλσβούργου που μπορεί να είναι ε, χρήσιμος για τους επιβάτες, όχι όμως για τη μεταφορά αγαθών. Πιστεύω ότι κάτι τέτοιο θα ήταν δυνατό να γίνει. τα κράτη-μέλη ήδη απειλούν να περικόψουν το προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τον ε, ε, ε, ε, μειωμένο προϋπολογισμό όμως κάθε κράτος μέλος θέλει να πετύχει τα περισσότερα. Χωρίς συγχρηματοδότηση δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Θα πρέπει όλοι να δούμε θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι όπου δεν υπάρχουν ε, χρήματα, ε, ακόμα και ο ε, αυτοκράτορας χάνει τα δικαιώματά του. Θα ήθελα πολύ να περιμένω να ακούσω τις απαντήσεις σας και ενδεχομένως να έρθω διμερώς σε επαφή μαζί σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κυρία Φάεν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους συντονιστές για τις λεπτομερείς τους εισηγήσεις. Επιτρέψτε μου να προωθήσω την προοπτική της Σλοβενίας συζήτηση. Απευθύνομαι στον κύριο Μπρίνκοστ. Χαίρομαι που υπογράμισε τη σημασία του έκτου, ε, της έκτης προτεραιότητας του έκτου ΠΠ. Στην ε, έκθεση αναφέρεται ότι η Σλοβενία έκανε μεγάλα βήματα σε ό,τι αφορά τη βελτίωση των σιδηροδρομικών υποδομών. Η πρόοδος αυτή όμως είναι κάπως αβέβαια. Υπάρχει ανάγκη καταρχάς να εξυγχρονιστούν οι σιδηροδρομικές δομές του διαδρόμου 5. Είναι ένας διάδρομος που αφορά ένα μεγάλο μέρος των μεταφορών εμπορευμάτων και στην Βόρειο Αδριατική. Περίπου το 60% της μεταφοράς εμπορευμάτων γίνεται σε αυτή την περιοχή, μέσω της Ουγγαρίας, μέσω της Αυστρίας. Συνεπώς αυτό τόσο διάδρομος είναι πάρα πολύ σημαντικός. Ο πέμπτος διάδρομος, το έκτο έργο συναντάται με τον διάδρομο 10 και είναι ένα σημαντικό σημείο συνάντησης. Ε, ένα σημείο που θα πρέπει να ενισχυθεί εν ώψη της διεύρυνσης στα Ανατολικά Βαλκάνια. Τις νέες χώρες μέλη μετά το 2004 δεν μπόρεσαν να να κερδίσουν το χαμένο χρόνο σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη. Το, δίκτυο, το, το δικό δίκτυο στη Σλοβενία έγινε κυρίως με τα δικά μας, ε, με τους δικούς μας ε, πόρους. Ε, και το μεγαλύτερο μέρος των πόρων διοχετεύτηκαν στο έργο υπαριθμών 6 για τους σιδηροδρόμους. Υπάρχει λοιπόν ανάγκη για μια συγχρηματοδότηση η οποία δεν τα λαμβάνει υπόψη μόνο τις χρηματοδοτήσεις ανά έργο, αλλά και το στοιχείο του πληθυσμού, τη βαρύτητα του πληθυσμού για τα μεμονωμένα έργα υποδομών. Ένα άλλα θέματα, προβλήματα που αφορούν τη συμφωνία του Τωρίνου μεταξύ της Ιταλίας και της Γαλλίας. Εάν δεν θα υπάρξει επιβεβαίωση αυτή τη συμφωνία με το τέλος του χρόνου, διατρέχει κινδύνους το έργο αυτό. Είστε αισιόδοξο. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί αυτή η συμφωνία, διακυβεύεται όλο το ε, σχέδιο, το όλο το έργο. Έχω την εντύπωση ότι μία αλλαγή των προτεραιοτήτων θα γίνει δεκτή ιδιαίτερα αρνητικά σε αυτό το μέρος της ε, ε Ευρώπης. Ο κύριος Σούζας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σήμερα το βράδυ η μεταφορά του Πατ Κόξ ε, με το αυγό και την κότα υπήρξε ιδιαίτερα επιτυχής. Θα ήθελα λοιπόν να του κάνω μια ερώτηση ανατρέχοντας και πάλι σε αυτή την, ε, μεταφορα... την παρομοίωση. Ε? Μπορώ να συνεχίσω. Ωραία. Ευχαριστώ. Το, η προτεραιότητα 1 γεννιέται ο αυγό στο Βερολίνο και θα έπρεπε να πεθάνει ο Σκότα στο Παλέρμο. Στην έκθεσή σας δεν γίνεται αναφορά στο θάνατο της Σκότας. Δεν γίνεται αναφορά στο Παλέρμο. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω συγκεκριμένα ποιοι είναι οι προβλεπόμενοι χρόνοι για την πραγματοποίηση, ποιο είναι το προβλεπόμενο κόστος, Ποια είναι η προβλεπόμενη χρηματοδότηση για να μπορέσει να γεννηθεί αυτή η κότα και ιδιαίτερα η γέφυρα στο στενό της Μεσίνης. Δεύτερη ερώτηση. Υπάρχει ένα σχέδιο Β για το Λιόν Τωρίνο γιατί είναι ανώφελο να αρνηθούμε την ύπαρξη προβλημάτων. Καλύτερα να ασχολούμεθα με εφαρμόσιμα προγράμματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ούγκας. Ο κύριος Κούν. Μην αναφέρετε το Στουτγάρ 21. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο και το είπαν αυτό και οι τέσσερις συντονιστές, να ασχοληθούμε με την οικονομική κατάσταση στον κόσμο. Από την από Ανατολή έρχονται πολλά αγαθά στην Ευρώπη και στη Μεσόγειο. Χρειαζόμαστε λοιπόν διάφορες δυνατότητες διανομής των προϊόντων αυτών. Δεν φτάνει να πούμε ότι ε, έχουμε διάφορα τούνελ ε, και όλα καταλήγουν σε ένα σημείο και δεν, δεν θα φτιάξουμε το τούνελ ε, του Μπρένερ. Θα πρέπει να υπάρχουν τρόποι τροφοδοσίας και της Ανατολικής Ευρώπης. Χρειαζόμαστε έναν λιμένα βαθέων υδάτων Ε, θα πρέπει να εξετάσουμε την κατάσταση στην ε, Τεριέστη, θα πρέπει να έχουμε ε, έναν λιμένα για κοντέινερ στο σημείο αυτό. Χρειαζόμαστε και το EMTS. Όσοι το θέλουν λένε ότι είναι πολύ χαμηλό το κόστος. Έχουμε όμως το Stuttgart 21 σαν μολόχ πάνω πολύ την υπόθεση. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε να, να ε, προχωρήσουν τα ε, θέματα αυτά με τον ίδιο τρόπο σε όλη τη Γερμανία και ε, θα πρέπει να εξετάσουμε αν η διαδρομή 1 ή η διαδρομή 22 θα προχωρήσει από το Βερολίνο Ροστόκ, αν θα προχωρήσει πιο βόρεια. Πάντως συμφωνώ απόλυτα. Εγώ πάντως είμαι υπέρ του Στουγάρτη 21. Um, Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ρίκε. Κύριε Πρόεδρε, θα σας μιλήσω για τη Στουτγκάρδη 21. Μολονότι οι γνώσεις μου για το, τους σιδηροδρόμους Αυστρίας, Γερμανίας έχουν προοδέσει πολύ. Θα θέλω να ευχαριστήσω τον Επίτροπο για την αφοσίωσή τους και για τη δουλειά που έκαναν και να κάνω το πρώτο ερώτημα. Ποιος ε, δεν εξεπλά... Πώς... Ε, ε, ποιος είναι αυτός που μπορεί να πει ότι δεν δοκίμασε να παραστήσει το Διευθυντή Ορχήστρα μπροστά στο ε, ραδιόφωνο Δηλαδή, Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε μία ή δύο παρατηρήσεις. πρώτη παρατήρηση είναι ότι όταν κοιτάμε τα έργα βλέπουμε ότι οι συντονιστές αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα. Αν κοιτάξετε τα πραγματικά μέσα που έχει στην ε, θέση της Ευρω... Ε, ε, διάθεση της Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε ένα δισεκατομμύρια ευρώ για, για το TNT. Βεβαίως δεν είναι πολύ μεγάλο ποσό. Δηλαδή διασχίζουμε, ε, κάνουμε ένα χιλιόμετρο το χρόνο, σε 55 χρόνια θα, θα τελειώσουμε. Η, όλη η πολιτική βρίσκεται στα χέρια των χωρών ή των περιφερειών μέσα και από, τα δικά μας κονδύλια, μέσα από τα διαφορετικά ταμεία. Συνεπώς το ερώτημα που τίθεται από το σύνολο των έργων είναι θα κάνουμε, θα προσποιηθούμε ότι ε, εμείς αποφασίζουμε την πολιτική ή θα προσπαθήσουμε να βρούμε τα μέσα για να το κάνουμε. Γιατί πραγματικά υπάρχουν διαφορές μεταξύ αυτού που νομίζουμε και του τρόπου που γίνονται τα πράγματα. Τώρα, το μέσα ένα συμβολικό θέμα που ξεπερνά τα όρια του συγκεκριμένου συστήματος ακόμα και αν μειωθούν τα προσκόμματα ακόμα και αν ανοίξει σύραγγα δεν θα πάει καλά το πράγμα, δεν υπάρχει εναρμόνιση, γιατί δεν υπάρχει ασφάλεια, γιατί δεν υπάρχει διαλειτουργικότητα ε, που να αφορά το υλικό και το προσωπικό και με έκπληξη άκουσα τον κύριο Βίνκ που έχει κάνει θαυμάσια δουλειά αλλά που μίλησε για, για το ΕΤΜΣ δίχως να αναφερθεί στην, στον Ευρωπαϊκό Φορέα Συνδυροδρόμων που είναι ε, στην ουσία το μόνο λειτουργικό στοιχείο που έχουμε στο παρελθόν το Κοινοβούλιο αρνήθηκε να δώσει 600.000 ευρώ στον φορέα αυτό Πραγματικά ε, είναι τρομερό, απίστευτο. Ε, υπάρχει πολιτική συνείδηση. Κύριε Βίκ, ε, όταν η Deutsche Bank σας λέει ότι θα δώσει ένα εκατομμύριο ευρώ το μήνα σε τέτοια μέσα, το κάνει. Το θέμα είναι ότι υπάρχει ένα πλεονέκτημα στο να διατηρηθεί αυτό το μονοπόλιο και η μη διαλειτουργικότητα είναι ο καλύτερος τρόπος για να γίνει. Θα ήθελα να τελειώσω την παρέμβασή μου. Δεν θα ήθελα να εξετάσω ε, τμήμα προς τμήμα ε, το Σαγκοτάρ, τη Μεσίνη, το Μπρένερο ε, και να συγκεντρώσω όλα τα προβλήματα που αφορούν την Αυστρία, τη Γερμανία. Θα ήθελα απλώς να πω ότι θα μπορούσαμε να έχουμε τη συνείδηση ότι εάν δεν πάρουμε πολιτικά την κατάσταση στα χέρια μας, εδώ οι συντονιστές κάνουν ό,τι μπορούν, αλλά θα συνεχίσουμε να βλέπουμε τις χώρες να διεξάγουν μια πολιτική ε, διακρατικών δικτύων. Ευχαριστώ. Κύριος Μπάχ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τους τέσσερις συντονιστές για τις ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις τους. Ήδη άκουσα τόσα από τους προλαλήσαντες που δεν έχω άλλες ερωτήσεις για τους ε, διαδρόμους. Έχω δύο συγκεκριμένες ερωτήσεις όμως ε, προς τον κύριο Βίνκ ε, όσον αφορά το RTMS. Είπε στην αρχή ότι ήδη σε 10 χώρες έχει εγκατασταθεί το σύστημα και ήθελα να ρωτήσω οι χώρες αυτές βρίσκονται στο ίδιο τεχνικό επίπεδο, το υψηλότερο και η δεύτερη μου ερώτηση ακολουθεί την ίδια κατεύθυνση. Γίνονται πολλές προσπάθειες ε, να εγκατασταθεί το RTMS, ε, αλλά με φόντο την ε, οικονομική κρίση μήπως έχουν ε, ε, καθυστερήσει τις επενδύσεις τους, μήπως δεν σκέφτονται καν να ε, προμηθευτούν τον εξοπλισμό αυτό και πώς μπορούμε να προχωρήσουμε, αναφέρατε κίνητρα, μπορείτε επίσης να ασκήσετε πίεση ή να θέσετε προθεσμίες, διότι τι νόημα έχει ακόμα και η καλύτερη υποδομή εάν το υλικό αυτό τελικά δεν χρησιμοποιείται. Μπορείτε επίσης να παράσχετε βοήθεια ώστε να μην υπάρχει χάσμα ανάμεσα στην ε, υποδομή και το ε, υλικό που ε, χρησιμοποιείται. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Κόχ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Κόξ. Δεν άκουσα τίποτα από εσά για το τέντι 1. Ε, το 16% των επενδύσεων έχει ολοκληρωθεί, όλες οι γέφυρες έχουν ολοκληρωθεί, όλες, όλες οι σύραγγες. Οι Γερμανοί πράσινοι ε, ζητάνε σταμάτημα διότι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι υποδομές αυτές ε, από τις οδικές μεταφορές. Γνωρίζετε άλλες περιπτώσεις όπου να καθυστερούν τόσο πολύ τα έργα και να αυξάνεται τόσο πολύ το κόστος τους. Ευχαριστώ η κυρία Βίλ. Ευχαριστώ. Κατά την εισήγηση του κυρίου ε, Μπάλας ε, μου έκανε ε, εντύπωση που άκουσα ότι ο άξονας Παρίσι-Βουκουρέστη σταματάει στην Στουτγάρδη ήθελα να ρωτήσω αν ο σταθμός της, του Γάρδης ε, λαμβάνει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Ακούσαμε πως όχι. Ε, αλλά ε, το βιβλίο που μας δώσατε είναι, συμβάλλει στην σύγχυση διότι δεν είναι πολύ σαφές αυτό που λέει. Αναφέρεται ο σταθμός Γκάρδη 21, αναφέρεται και ο υπόγειος ε, σταθμός. Η κυρία Μέρκελ επένεσε το έργο αυτό και είπε μάλιστα ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αποφασίσει την ε, κατασκευή του σταθμού αυτού. Ο σταθμός της σε βρίσκεται σε ε, ένα φαράγγι, σε μια λεκάνη και είναι ε, πολύ σημαντικό έργο το ότι έχουν, πετύχει ένα, το ότι έχουν βρει ένα σχέδιο όπου να, που να μπορεί να προσεγγιστεί χωρίς ε, γέφυρες, χωρίς τούνελ κλπ. Υπόθηκε ότι οι τοπικές μεταφορές και οι μετακινήσεις αγαθών δεν μπορούν να υποφεληθούν από το έργο αυτό. Μήπως μπορούμε να δαπανίσουμε καλύτερα τα σχετικά χρήματα. Ευχαριστώ στο τέλος του καταλόγου. Τέλος, ε, ο κύριος Κάτσης, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριοι συντονιστές, καταρχάς εκτιμώ ιδιαίτερα το στόχο σας ε, να προσπαθήσετε να κάνετε μια συζήτηση επί της ουσίας και να μας ενημερώσετε και να μας πληροφορήσετε για τι συμβαίνει. Το πιο σημαντικό είναι ότι τα μέσα για να επενδύσουμε στις υποδομές ε, των σιδηροδρόμων είναι περιορισμένα και έχουμε ανάγκη πολύ περισσότερα κονδύλια. Ε, τα χρήματα τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας δε, δεν ξέρουμε να τα χρησιμοποιήσουμε με το σωστό τρόπο. Δεν καταφέρνουμε να τα απορροφήσουμε αυτά τα κονδύλια και δεν υπάρχει ούτε ένα πρόγραμμα το οποίο να μην παρουσιάζει καθυστέρηση. Αυτό είναι παράδοξο αν λάβει υπόψη κανείς ε, τις πολιτικές μας προτεραιότητες. Οι επενδύσεις όταν κατασκευάζεται μια συγκεκριμένη υποδομή Όταν ενημερώνονται οι πολίτες, ε, οι πολίτε τα οικειοποιούνται αυτά τα προγράμματα, τα χαιρετίζουν με ενθουσιασμό και περιμένουν πότε θα υλοποιηθούν. Εγώ θα ήθελα να σα ρωτήσω το εξή. Έχετε ένα εναλλακτικό σχέδιο, ένα εφεδρικό σχέδιο, δεν λέω για ένα εναλλακτικό διάδρομο, αλλά έστω ότι ε, δεν υλοποιείται. Έχετε ένα εφεδρικό σχέδιο, ένα νέο προσανατολισμό των μέσων που δεν απορροφήθηκαν ε, προς τα, ε, τους διαδρόμους που λειτουργούν για να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε μια καλή δυναμική ώστε να μπορέσουμε και εμεί, ω Ευρωπαϊκό Θεσμικό Όργανο να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε ε, κατάλληλα τα κονδύλια που ε, κατανέμουμε. Εγώ δεν είμαι η Δήμων περί των οικονομικών, αλλά υπάρχουν συνάδελφοι που μπορούν να σα εξηγήσουν τι γίνεται με τα κονδύλια τα οποία δεν απορροφούνται κάθε χρόνο. δεν μπορούμε να συγκεκριμενοποιήσουμε τα προγράμματα, τίνουμε να καθυστερούμε τις προθεσμίες και να τις αναβάλουμε συνεχώς ε, για διάφορα προγράμματα. Ακόμα και στη χώρα μας ε, που λέγεται ότι δεν έχουμε τα οικονομικά μέσα για να απορροφήσουμε ευρωπαϊκά κονδύλια, είναι αλήθεια ότι πρέπει να είμαστε όλοι πολύ πιο ευέλικτοι για την απορρόφηση των κονδυλίων και για τον επαναπροσανατολισμό τους προς τα προγράμματα τα οποία θα μας δώσουν την απαραίτητη δυναμική. Πρέπει να το κάνουμε, υποχρεούμεθα να το κάνουμε, διότι αν δεν σεβαστούμε την αρχή της καλής ε, οικονομικής διακυβέρνησης, δεν θα μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε στον καλύτερο δυνατό βαθμό τα κονδύλια μας. Και προς το παρόν η πραγματικότητα αποδεικνύει ότι δεν καταφέραμε να διαχειριστούμε σωστά τα κονδύλια. Πριν δώσω το λόγο στους συντονιστές ε, και ακούσω τις δικές τους ερωτήσεις, απαντήσεις, συγγνώμη, ε, να πω κάτι εγώ. Δεν είχα σκοπό να μιλήσω, αλλά ο κύριος Ρίκε είπε κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και σωστό και νομίζω ότι αυτό είναι το θέμα του RTMS. Κάτε με, το RTMS είναι το κλειδί που ξεκλειδώνει το κλειδί της, ε, την πόρτα της διαλειτουργικότητας. Αν δεν βρούμε το σωστό κλειδί, η πόρτα θα μείνει εφτασφράγιστη για σας. Ανεξάρτητα από τι είπαμε, μπορούμε να χαράσουμε όσε γραμμέ θέλετε στου χάρτε. Είμαστε πάρα πολύ καλοί σε αυτού του χάρτε. Πολύ συχνά λέω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, λέω μην ετοιμάστε χάρτη, γιατί οι πολιτικοί του λατρεύουν του χάρτε. Αλλά το θέμα είναι τι γίνεται στην ουσία. Και το βασικό για μένα, συνάδελφοι, ε, είναι η χρηματοδότηση ε, τα κονδύλια και οι προτεραιότητες. Θα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητες σε αυτά που θεωρούμε σημαντικά για το τμήμα των Ευρωπαϊκών Σιδηροδρόμων και για μένα δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το ERTMS, διότι όπως σας είπα αυτό είναι το κλειδί που ξεκλειδώνει την πόρτα. Είναι το στοιχείο που καλύπτει, αν θέλετε, το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο ένα τμήμα της. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να το σκεφτούμε λίγο αυτό Ιδίω επειδή έχουμε περίοδο λιτότητας ε, δεν μας περισσεύουν ε, και χρήματα και νομίζω ότι ε, είχε δίκιο ο κύριο Ρίκε όταν το ανέφερε. Χωρίς αυτό το κλειδί η πόρτα της διαλειτουργικότητα των σιδηροδρόμων θα παραμείνει ερμητικά κλειστή. Ωραία, να δώσω το λόγο στους συντονιστές με την ίδια σειρά που τους αναδείξω και προγραμμένος. Ο καθένας έχει από ένα-δύο πράγματα να μας αναμασίσει επειδή οι συνάδελφοι έθεσαν πάρα πολλές ερωτήσεις και έκαναν πάρα πολλές παρατηρήσεις, αυτό δεν σημαίνει ότι εσείς έχετε απεριόριστο χρόνο στη διάθεσή σας. Ήθελα απλώς να σας το πω αυτό. Θα ξεκινήσω από εσά κύριε Κόξ, λοιπόν. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη για τα σχόλιά τους και θα ήθελα να απαντήσω στα ερωτήματα που μου τέθησαν. Κύριε Κατσάνο, συμφωνώ μαζί σας. Έχουμε μάθει από το παρελθόν βεβαίως και θα πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές αλλά και αισιόδοξοι για το μέλλον. Έχετε δίκιο για το θέμα της χρηματοδότησης, δεν θα το θίξω. Σε ό,τι αφορά το θέμα της συγχρηματοδότησης, οι προσδοκίες δεν νομίζω ότι θα μειωθούν με το πέρασμα του χρόνου. Πρόκειται για ένα στρατηγικό θέμα. Συμφωνώ μαζί σας, οι συντονιστές δίχως άλλο έχουν ένα ρόλο να διαδραματίσουν σε ό,τι αφορά τις τοπικές αναποτελεσματικότητες θα συμβάλλουν δίχως άλλο στην ανέβρεση λύσεων. Αυτό είναι ένα ρόλος που αποδεχόμαστε για τον εαυτό μα. Η κυρία Λισέντερ έθεσε ερωτήματα για την ενδιάμεση έκθεση. Έχετε δίκιο όταν λέτε ότι κατεγράφησαν σημαντικές ε, καθυστερήσεις ακόμα και σε επίπεδο προγραμματισμού, για να μην μιλήσουμε για τις κατασκευές. Υπάρχει ένα πρόβλημα στο δυτικό στον νότιο ε, άξονα και θα πρέπει να υπάρξει, να περάσουμε στη φάση σχεδιασμού και κατασκευής. Θα πρέπει να πω ότι τα όσα έχουν γίνει στο Πόντε Γκαρντένα και στην Φορτέτσα και, στην, ε, και στο Μπολτζάνο βρίσκεται αρκετά πιο μπροστά και είναι πιθανό κατά την άποψή μου να χρησιμοποιήσει τα περιθώρια ελαστικότητας τα οποία αναφέρθηκε ο Επίτροπος. Δηλαδή θα υπάρξουν πολιτικοί και οικονομικοί και κοινωνικοί όροι που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας μέχρι το 2013. Πιστεύω ότι θα μπορέσουν τα σημεία αυτά να πάρουν ε, να, να εκμεταλλευτούν αυτό το περιθώριο ε, λαστικότητας. Σε ό,τι αφορά τα άλλα στοιχεία, δηλαδή την παράκαψη του Τρέντο και την πρόσβαση στη Βερόνα, με βάση τις λεπτομερείς πληροφορίες που είχα, έχω την εντύπωση ότι σε ό,τι αφορά τη φάση της σύλληψης βρίσκονται αρκετά πίσω και υπάρχει ο κίνδυνος εξετάζοντας την ενδιάμεση έκθεση ότι τα κονδύλια που έχουν μπει στην άκρη για τη χρηματοδότηση ενδεχομένω θα χαθούν. Θα ήθελα να τονίσω αυτό που είπε ο αρμόδιος επίτροπος. Οποιοδήποτε πρόγραμμα, ε, σχέδιο είναι βιώσι, έργο είναι βιώσιμο στο μέλλον θα μπορούσε να επανέλθει στον επόμενο γύρο του προπολογισμού. Δεν είναι ότι κάτι χάνεται διαπαντός σε ό,τι αφορά την χρήση των κονδυλίων τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή ενδεχομένως ε, ορισμένα έργα θα ενταχθούν σε ένα μετέπειτα χρονοδιάγραμμα. Υπάρχει λοιπόν μια διαφοροποίηση εδώ να πιστεύω ότι θα επιτευχθεί η πραγματική πρόοδο. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι το θέμα αυτό ετέθη αρκετέ φορέ κατά τη διάρκεια των ε, ανταλλαγή απόψεων ε, που είχαμε, αν μπορούμε να τις επισκεφτούμε τις διάφορες αρχές κτλ. Στην Ιταλία ε, έχουν καταβληθεί πάρα πολλές προσπάθειες για να δοθεί μια απάντηση στις επικρίσεις που έχουν γίνει από πλευράς του ελεκτικού συνεδρίου και προσπάθησαν να σταθούν στο ύψος των απαιτήσεων του ελεκτικού συνεδρίου. Όλα αυτά θα μπορούσαν να ε, που θα μπορούσαν να θεωρηθούν υποδομές απέτησαν χρόνο και πιστεύω ότι αποτελεί ένα μήνυμα καλής θέληση από πλευρά των Ιταλικών αρχών. Βεβαίω, σας είπα ότι θα υπάρξει μια καθυστέρηση σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Η κυρία Μάισεν ερέθεσε το ερώτημα για τη Γερμανία και συγκεκριμένα για τον Βόρειο Άξονα όλα αυτά συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση, αλλά θα ήθελα να αναφερθώ στην πρόοδο που επετέφθη. Η... Όλες αυτές ε, οι υπηρεσίες ε, υπάρχουν. Νομίζω ότι οι παραδόσεις ε, θα γίνουν σωστά 2015-2017 ενώ άλλα έργα θα τελειώσουν το 15. Ο κύριος Κρέιμερ έθεσε το ερώτημα του κατά πόσο θα γίνουν σεβαστά αυτά τα χρονοδιαγράμματα. Ακούστε, εγώ σας λέω όσα μου είπαν και τα άκουσα καλή την πίστη. Ο Υπουργό Άντα μου είπε ότι αυτά τα τμήματα θα παραδοθούν έγκαιρα. Και οι υπεύθυνοι στο Υπουργείο Υποδομών μου είπαν ότι όντω θα παραδοθούν έγκαιρα. Όταν τίθεται το ερώτημα των, ε, του άξονα μόναχο αυστριακά σύνορα, εδώ υπάρχει ένας κίνδυνος να υπάρξει μία παρέκκληση μολονότι δεν, δεν θα πρέπει να απομαγνηθούμε τόσο πολύ ε, έτσι ώστε να φτάσουμε σε ένα κρίσιμο σημείο. Ε, Βεβαίω το να υπάρχει η σύραγγα χωρί οδού ε, πρόσβαση είναι σαν να έχει κανεί μια Ιρλανδέζικη μπαμπ που να μην σερβίρει μπύρα. Ε, στο χρονοδιάγραμμα στη Γερμανία. Σε ό,τι αφορά τη γέφυρα τη μεσίνη. Ε, ε, εγώ εστίασα την προσοχή μου στην, στο νότιο άξονα. Είπατε ότι έχω μία λαθασμένη αντίληψη της πραγματικότητας. Να περιμένουμε. Είτε εσείς έχετε δίκιο, είτε εγώ. Ε, του, του, χρόνου θα έχουμε να κάνουμε με τη Φορτέτσα και το Ινσπρουκ. Ε, θα δούμε τι θα γίνει. Βεβαίως ε, δεν θα ξεκινήσει όλο μαζί και πραγματικά μετά από ένα χρόνο, αν έρθω εδώ και σας μιλήσω και σας πω ότι αυτό δεν έχει γίνει, αυτό θα είναι πηγή μεγάλης απογοήτευση. Και σε ό,τι αφορά το ρόστο, το θέμα του Core Network δεν συμπεριλαμβάνεται στο διάμεση έκθεση. Είμαι πεπισμένο όταν ακούω αυτά. Κύριε Κούρα, αναφερθήκατε στο θέμα των Αδριατικών λιμένων. Έγινε μια θαυμάσια παρουσίαση στο Βερολίνο από τον κύριο Κάστα που περιέγραψε τις ε, δυνατότητα με ε, χρήσης αυτών των οδών για την ε, διαμετακόμιση στην Ευρώπη. Αυτοί που λένε ότι στην ε, ε, Ελβετία θα φτάσουμε στο ανώτατο σημείο του δυναμικού, νομίζω ότι παρουσιάζουν ένα ψευδές επιχείρημα. Ε, ε το θέμα είναι πώς θα συνδεθούμε με αυτό το core network. Υπάρχουν ε, σημαντικές, ε, σημαντικά θέματα που θα πρέπει να εξεταστούν. Κυρία Μπέρνερ έθεσε το ερώτημα για την Ιταλία και τους διάφορε θύμες που υπάρχουν. Στην Ιταλία είδα ότι έχει καταγραφεί πραγματική πρόοδος ακόμα και σε επίπεδο γραφειοκρατίας. Υπάρχει βούληση και δίχως άλλο αυτό θα διευκολύνει τα πράγματα και θα μπορέσουμε να παραδώσουμε ένα μέρος του έργου. θα γίνει και μια συνάντηση στις 19 Νοεμβρίου. Σε ό,τι αφορά τις δυσκολίες με το ε, ανάγλυφο, εγώ δεν είμαι ειδικό. Μίλησα με τον κύριο Κόρναλ Μπέρκμαϊστερ, όπως γνωρίζετε, είναι επικεφαλής του BBTSC και έκαν, ε, ήδη έχουν ανοίξει αρκετές σύραγγες συμπεριλαμβάνοντας και ε, ε, ε, ορισμένα ρήγματα στην περιοχή γύρω από την Αδριατική. Ξέρουν τι κάνουν και ξέρουν και πώς θα το παραδώσουν. Κυρία Λίχτεμπεργκερ, σχετικά με το θέμα της πρόσβασης από το, το Νότο. Αυτό είναι ένα θέμα που θα πρέπει να μας απασχολήσει. Το θέμα της χρηματοδότησης μέσω της Eurovignette του cross-financing της χρηματοδότησης από το χερσαίο στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Νομίζω λοιπόν ότι αυτά θα πρέπει να τα εξετάσουμε περαιτέρω. Στην Αυστρία θα πρέπει να πάρουμε τα ήδη υπάρχοντα παρόλο που πολλά ακόμα μπορούν να γίνουν. Δίχως άλλο θα σας κρατήσω ενήμερου στην... Σε ό,τι αφορά το θέμα της ε, κότας και του αυγού και το Παλέρμο, τι να σας πω, δεν είχα λεπτομερείς συζητήσεις μέχρι τώρα σε ό,τι αφορά το στενό της Μεσίνας. Ε, συμφωνώ με το σχόλιο που έκανε, κάντε για το πρόεδρο του Μέσα. Κύριε Κάρτον, θέσατε το ερώτημα για τον προϋπολογισμό. Δεν νομίζω ότι ως συντονιστές θεωρήσαμε κάτι για το πρόγραμμα Β. Θα μπορούσα να σας πω ότι πέρσι δούλεψα εθελοντικά και εις βάρος του προσωπικού μου χρόνου ε, για το θέμα αυτό και με απασχόλησε το θέμα των προοπτικών 2007-2013. Ε, και εάν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα αυτό δεν φορά το μεταφορές αποφάσισαν να ξεφύγουν από τις δεσμεύσεις τους δηλαδή ε, ε, σε ό,τι αφορά τον καθορισμό των προτεραιοτήτων κοιτάξτε οι συντονιστές δεν είναι πλέον κατάλληλοι να το κάνουν uh, uh, Ευχαριστώ πολύ Πάτ θα ήθελα να πω ότι ε, μια Ιρλανδική pub χωρίς μπύρα θα ήταν ε, λόγος για κοινωνική ε, διαμαρτυρία. Ο κύριος Πάλλας. Κύριε Κράμερ. Δεν ανέφερα καθόλου τη Στουτγάρδη 21, διότι δεν είναι ευρωπαϊκό έργο. Αυτό μπορώ να το ε, ξαναεπιβεβαιώσω, ε, το είπε αυτό και ο ίδιος ο Επίτροπος. Στην Γερμανία μπορεί να υπάρχουν παρανοήσεις, εμείς όμως ε, και εγώ και εσείς και όλοι οι άλλοι που βρίσκονται εδώ το έχουμε ήδη αναφέρει επανειλημμένα. Το γνωρίζουμε. Η Ευρώπη χτίζει δίκτυα, γραμμές, όχι σταθμούς. Επικροτούμε την κατασκευή σταθμών Ήδη το έκανα σήμερα. Ανέφερα τον νέο σταθμό ε, ε της ε, του ε, Σεντ Πέλτεν. Δεν αναφέρθηκα στο Στρασβούργο. Αλλά και στο Στρασβούργο έχει γίνει εξαιρετική δουλειά κατασκευής του σταθμού. Όλα αυτά είναι σημαντικά. Πρέπει να είναι απόλυτα σαφές όμως ποιος χρηματοδοτεί τι. Τι χρηματοδοτούν οι χώρες, οι περιφέρειες, ε, οι, οι πόλεις. Είναι αξιοπρόσεκτο ότι τα τελευταία χρόνια δεν, είχαμε, δεν είδαμε σημαντικές δυσκολίες στη Στουτγάρδη. Γιατί ε, έχουν ξεσπάσει τώρα οι διαμαρτυρίες αυτές εσύ σίγουρα το γνωρίζετε καλύτερα από μένα. Εγώ μπορώ μόνο να υποθέσω ότι αυτό συνδέεται με το ξεκίνημα των κατασκευαστικών εργασιών. Έτσι, ο κόσμος βλέπει με τα ίδια του τα μάτια ότι έχει ξεκινήσει η δουλειά. Τώρα ε, εξετάζεται η αύξηση του κόστους και έχει αυξηθεί σημαντικά το κόστος. Στην αρχή η εκτίμηση ήταν 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Σήμερα μιλάμε για 7 δισεκατομμύρια. Αύξηση 50%. Ως ιδιώτες δεν είναι βέβαιο ότι θα αγοράσουμε το ίδιο προϊόν ε, μετά από αύξηση τιμής κατά 50%. Ε, μπορεί να ήταν αποδεκτή η τιμή κάτω των 5 δισεκατομμυρίων ε, ενώ η παρούσα τιμή δεν, είναι, δεν ξέρω αλλά υποθέτω ότι αυτό συμβαίνει ότι η τιμή έχει παίξει κάποιο ρόλο. Η πολιτική κατάσταση έχει επίσης αλλάξει και ας μην ξεχνάμε και την γενική οικονομική κατάσταση, τα προβλήματα ε, τα δημοσιονομικά σε όλα τα κράτη-μέλη και στη Γερμανία. Έχουμε λοιπόν από τη μία αύξηση της τιμής, από την άλλη ε, οικονομικές δυσκολίες που οδηγούν στην παρούσα κατάσταση. Η λύση θα πρέπει να βρεθεί στην Γερμανία, στην Βάδη Βιρτεμβέργη και στην ίδια την πόλη της Στουτγάρδης. Και η λύση θα πρέπει να είναι πολιτική, οικονομική και τεχνική η Στουτγάρδη έχει πολύ έντονη τοπική κίνηση. Ε, πολλοί κόσμος ε, πηγαίνει στη Στουτγάρδη να δουλέψει και μετά επιστρέφει στο σπίτι του. Οι διεθνείς ε, μεταφορές ίσως παίζουν μικρότερο ρόλο. Αυτό είναι σημαντικό για όλους τους άλλους. Ε, πολλοί φίλοι με έχουν ερωτήσει πότε θα λειτουργήσει αυτός ο υπέροχος σιδηρόδρομος πότε θα μπορούμε από την Βαρσοβία, το Βουκουρέστι και τη Βουδαπέστη να ε, πετάμε στο, στην Γερμανία για να πάρουμε κατόπιν ένα ε, ε, υπερταχή τρένο για το, το Στρασβούργο. Πολλοί συνάδελφοι με ρώτησαν. Επίσης, τους ενδιαφέρει η σύνδεση με το αερο αεροδρόμιο. Είναι λοιπόν πολύ σημαντική η σύνδεση αφενός με το αεροδρόμιο και από την άλλη να υπάρχουν διεθνείς υπερταχείες αμαξοστοιχίες από το αεροδρόμιο. Και τα δύο αυτά είναι σημαντικά, είναι δύο διαφορετικές πτυχές όμως. στην ε, ευρύτερη περιοχή είναι πρόβλημα ε, ο σταθμός του 21. Ε, το πρόβλημα για μένα είναι η ίδια Στουτγάρδη και η διαδρομή. Αυτό είναι αδιέξοδο. Ανέφερα τα προτερήματα του σύνδεσμου Στουτγάρδη-Παρίσι, το ότι μπορεί κανείς να φτάσει μέσα σε τέσσερις ώρες στο Παρίσι. Υπάρχει και σημαντική βελτίωση στην Αυστρία και στην Βαβαρία Ε, υπολογίζουμε στη, μεταφορά, στη μετακίνηση αγαθών παράλληλα με τη μεταφορά επιβατών. Η διαδρομή από το Μόναχο θα περνάει από το Μίλντορφ και όχι από το Ρόζενχάιμ όπως ε, συνέβαινε παραδοσιακά για τους επιβάτες. Αυτό είναι χρήσιμο και για την ε, αγαθών. Οι τέσσερις συντονιστές ε, συναντήσαμε τον κύριο Ράμζαουερ στις 4 ε, Σεπτεμβρίου στον, στο Βερολίνο. Εγώ ίδιος θα πάω στο Μόναχο στις 5 Νοεμβρίου ώστε με να συνεννοηθώ στην Βαβαρία για όλα τα προγράμματα. Συνεχίζουμε δηλαδή να ασχολούμαστε με το θέμα. Τι άλλο είχα να πω. Και εντός της Γερμανίας θα πρέπει να ξεκαθαριστούν τα διάφορα συμφέροντα. Κατόπιν έρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειαζόμαστε λοιπόν συνεννόηση, συμφωνία ε, μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών. Κατόπιν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στη χρηματοδότηση. Εγώ πολύ ευχαρίστως θα χρηματοδοτήσω έργα μεταξύ κρατών μελών, όχι όμως εντός των κρατών μελών. Όσον αφορά το RTMS, ε, με ρωτήσατε, αλλά αυτό είναι αρμοδιότητα του συναδέλφου. Όχι, συγκεκριμένα ρώτησα τι βελτίωση θα επιφέρουν οι συγκεκριμένες διαδρομές. Ε, όσον αφορά την ε, εξοικονόμηση εκπομπών ε, διοξείδου του άνθρακα κλπ. Ναι, και εγώ αναφέρθηκα στο έλλειμμα στις μεταφορές αγαθών. Η απάντησή μου είναι ότι τώρα μόλις ξαναβλέπω το θέμα θα το εξετάσω και όπως και στο παρελθόν θα έρθω σε άμεση επαφή μαζί σας. Σας το υπόσχομαι ότι πριν το τέλος Νοεμβρίου θα έχετε συγκεκριμένη απάντηση στα ερωτήματά σας. Σήμερα δεν μπορώ να απαντήσω. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπριγχορστ έχετε το λόγο και όπως μάλλον μαντέψατε μας αρέσει η Σλοβενία. Ελπίζουμε λοιπόν να μην την παραλείψετε. Ναι, κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμο το γεγονός ότι ο Επίτροπος αναφέρθηκε στη μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση. Θεωρώ ότι πολλά από τα ερωτήματα επικεντρώνονται γύρω από αυτό το θέμα. Η πρώτη ερώτηση ήταν ε, «Είστε ικανοποιημένο, είπε η κυρία Γιάλα Σέντερ. Ναι, είμαι πολύ ικανοποιημένο, διότι θεωρώ ότι πλησιάζει η ώρα της αλήθειας. Ε, ο συνάδελφος έκανε την ίδια παρατηρήση με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή, τα κράτη-μέλη θα διοικούν την Ευρώπη ή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, που τώρα αποκαλείται Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει ακόμα κάποιο ρόλο να διαδραματίσει. Και παραδόξως, κατά κάποιο στρατηγικό τρόπο, η μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση θα υπηρετήσει την ευρωπαϊκή διάσταση. Και θα την υπηρετήσει με ποιο τρόπο. Διότι επειδή εγώ ήμουν μέλο ε, του συγκεκριμένου φορέα εδώ και κάποια χρόνια, Συνεχώ αναζητούμε νέα χρήματα και νέα επιρροή. Και είναι ευπρόσδεκτη αυτή η αλλαγή. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει. Και εδώ μιλάω και λίγο εκτό αρμοδιοτήτων, μπορεί να είμαι και επικίνδυνο, ε, μπορεί να πρέπει να κάνω και χαρακτήρι μετά από αυτά που θα σα πω. Αλλά νομίζω ότι αυτό που έχει σημασία είναι ότι πράγματι πρέπει να κάνουμε επιλογέ. Και το να κάνει κάποιε επιλογέ σημαίνει ότι θα έχει και τα μέσα και το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απλώς υπηρετεί τα κράτη-μέλη αλλά έχει να διαδραματίσει και κάποιο δικό της ρόλο. Τι σημαίνει με αναθεώρηση. Σημαίνει ότι από το 2030 μέχρι το 2050 ε, τα κράτη-μέλη θα είναι, συγγνώμη, 2013 ε, μέχρι το 2015 τα κράτη-μέλη θα είναι υπεύθυνοι και για τις επιλογές τους και θα πρέπει να κάνουν συγκεκριμένε επιλογές. Και έχουμε και την ερώτηση του κυρίου Κράμερ, ο οποίος μου είπε ότι μου εύχεται κάθε επιτυχία και ε, κατά πόσον πιστεύω ότι φτάσαμε στην ώρα της αλήθειας. Ναι, φτάσαμε στην ώρα της αλήθειας. Δεν μπορώ να προβλέψω τι θα κάνουν η γαλλική και η ιταλική κυβέρνηση με τη συνθήκη. Εγώ έχω τις απόψεις μου, ε, ε τις γνωρίζουν, δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνω εγώ τι έχω ήδη ξαναπεί. Αλλά ω συντονιστή και με τη δική σας ψήφο εμπιστοσύνη, αυτό που έχει σημασία είναι ότι είναι στρατηγικού συμφέροντος και για τους Γάλλους και για τους Ιταλούς. Και εάν δεν συμβεί, και θα επανέλθω σε αυτό ε, σε ένα λεπτό, η υπόλοιπη γραμμή θα είναι άχρηστη. Ελπίζω να μην είναι πρόκληση προς τον κύριο Κράμερα, αλλά δεν θα χρησιμοποιήσω το θέμα εδώ, αλλά το θέμα είναι ότι η ευθυγράμμιση από ιταλικής πλευράς χρήζει σαφήνειας. Αν δεν υπάρξει συμφωνία για τη χρηματοδότηση λοιπόν, θα αποδεσμευτούν κάποια κονδύλια και θα τα πάρουν άλλοι φυσικά. Μπορεί να γίνομαι λίγο κουραστικός εδώ, αλλά η μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση είναι και ένας μηχανισμός ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών μελών και πρέπει να έχουμε και το θάρρος της γνώμης μας. Είναι ένα μέσο ανταγωνισμού, διότι αν κάποια κράτη-μέλη δεν είναι έτοιμα, εγώ θα χάσω τη δουλειά μου και έχει σημασία για μένα, αλλά τα χρήματα θα πάνε αλλού. Ελπίζω να είναι σαφές αυτό. Και αυτό το στοιχείο νομίζω είναι ένα νέο στοιχείο το οποίο εμφανίζεται για πρώτη φορά. Το είπα και στην εισαγωγή μου ε, συντομία. Αν αυτή η γραμμή μεταξύ Σλοβενίας και Ιταλίας συμφωνηθεί, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είναι πλήρης εταίρος. Στο αρχικό κείμενο έλεγε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είναι παρατηρητής και με την έγκριση του Επιτρόπου Κάλλας ε, είπα ότι είναι λίγο παράδειξο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συγχρηματοδοτεί και να είναι παρατηρητής. Και αυτή είναι και απάντηση προς τον κύριο Ρίκε. Δεν είμαστε ένας διακυβερνητικός οργανισμός και το ίδιο ισχύει αν μετά το τωρινό και την χρηματοδότηση ε, που θα συμφωνηθεί, και αυτό δεν μπορώ να το προβλέψω, δεν είμαι μάντης, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συμμετέχει πλήρως υπάρχει το LTF που είναι η προκαταρκτική δομή, οι Γάλλοι και οι Ιταλοί και εμεί θα κάτσουμε και θα πούμε κατά πόσο μα αρέσει όχι. Κάποιοι λέμε ναι, κάποιοι λέμε ότι υπάρχουν δυσκολίε, αλλά στο μέλλον δεν θα γίνεται έτσι. Η έλλειψη πόρων θα είναι και ένα μέσο για να κατευθύνουμε τα κονδύλια τελικώς. Και αν δεν είναι διατεθειμένος, δεν πειράζει τι να κάνουμε, πάμε στον επόμενο. Ε, ο Λιόν ε, το Ρήνο θα είναι στρατηγική διάσταση διότι ε, δεν μπορεί να μην έχετε τη Λιόν που είναι η δεύτερη πόλη της Γαλλίας ενωμένη με το Τωρίνο. Καταλαβαίνετε ότι είναι κλειδί αυτός ο κόμβος είναι στρατηγική διάσταση, διότι Ανατολή Δύση είναι στρατηγική διάσταση. Το κατά πόσο θα συμβεί ενώ εγώ είμαι εν ζωή, ελπίζω να συμβεί και εξαρτάται από την καλή βούληση του καθενό και την εφευρετικότητα των κρατών μελών. Ζητώ συγγνώμη που μακρηγόρησα για το σημείο αυτό, αλλά να συνεχίσω τώρα με τη Σλοβενία. Ναι, έχετε δίκιο. Όπω και στη δεκαετία του 80 που εγώ ήμουν υπεύθυνο για την ενεργειακή πολιτική στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ισπανία έλεγε γιατί να μην έχουμε ένα αυτοκινητόδρομο μεταξύ Μαδρίτης και Βαρκελόνης ή Μαδρίτης προς το βορρά. Εσείς κάνατε κακό στο περιβάλλον σε βορρά, γιατί να μην έχουμε κι εμείς ένα αυτοκινητόδρομο. Συμφωνώ μαζί σας. Υπήρχε ε, κάποια στιγμή ένα ταξίδι στο οποίο εγώ έκανα ένα ταξίδι με ελικόπτερο σε όλη τη χώρα. Ευτυχώς οι συνθήκες επιτρέπουν σε δύο ώρες να δούμε με ελικόπτερο τη χώρα και είναι εκπληκτικό αυτό που έγινε στους δρόμους. Μαδρίτη Βαρκελόνη, ναι. Δεν έχει σχέση με εσά τώρα αυτό κύριε Κάντσα. Άλλη ερώτηση είναι ο κύριος Φλάτζης ήταν σημαντικός παράγων, διότι είπε ότι πλέον πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα και από αυτοκινητόδρομο να πάμε σε σιδηρόδρομο. Δυστυχώ δεν μπορούμε να ξαναφτιάξουμε την ιστορία. Εσεί είστε νέα γενιά και για μένα η Σλοβενία είναι εξίσου σημαντική με την Ολλανδία και με οποιαδήποτε άλλη χώρα. Και δεν θα είμαι εγώ αυτό που θα κρίνω ε, εάν ε, πρέπει να τα αριθμίσουμε αυτά στι υποδομέ. Αλλά μπορείτε κι εσεί να βοηθήσετε. Και να βοηθήσετε να ε, ε, χαθεί και όλη αυτή η απειλή του παρελθόντος. Έχω διαβάσει τα πάντα για την Τεργέστη και το πρόβλημα και τη σχέση μεταξύ Σλοβενίας και Τεργέστης αλλά να θυμάστε ότι στο μέλλον και νομίζω ότι και ο κύριος Κούμος έθεσε την ίδια ερώτηση ο κύριος Κούν στο μέλλον μία, σχε... Ε, μία σύνδεση με την Τεργέστη είναι ευρωπαϊκή σημασία. Στο να εκτρέψουμε ε, τη γραμμή από την Τεργέστη στην ε, Βάρτσα είναι πολύ σημαντικό. Καταλαβαίνω ότι είναι θέμα ιστορίας, αλλά τώρα υπάρχει η συμφωνία μεταξύ των πέντε βόρειων βασικών ε, στιγμών και έγινε και ένα σχόλιο για την Κίνα. Ναι, οι Κινέζοι δεν ξέρουν ούτε καν που είναι η Τεργέστρη, ούτε που είναι το Κόπερ. Το ίδιο θα έλεγα αν μιλούσε και για την Αμβέρσα. Χαίρομαι που δεν είναι εδώ, κυρία Πάτ. Αλλά οι Ολλανδοί αναφέρονται στην Αμβέρσα και στο Ρότερνταμ λες και βρίσκονται σε δύο διαφορετικούς πλανήτες. Ευτυχώς αλλάζουν λίγο τα πράγματα, αλλά το κόπερ και η ταιριαστή είναι 5 χιλιόμετρα απόσταση. Και δεν επιτρέπεται να περάσει ένα σιδηρόδρομο από εκεί και αρνούμαστε να κάνουμε μια σωστή γραμμή. Ελπίζω να σα πείσω και να υπάρχει μια νέα ε, αποδοχή από τη Σλοβενία και από την Τεργέστη για να προχωρήσει το θέμα. Μια τελευταία παρατήρηση. Το θέμα του εφεδρικού σχεδίου. Νομίζω ότι ο κύριος Κόξ ε, το σχολίασε. Δεν το σχολιάζουμε εμείς, δεν το εφαρμόζουμε. Εμείς είμαστε συντονιστέ. Αλλά να σας πω κάτι από την επιχειρηματική μου πείρα που απέκτησα πριν από πολλά χρόνια. Γιατί πετυχαίνουν οι Ιαπωνέζοι σε τομείς στους οποίους οι Ευρωπαίοι πολλές φορές έχουν αποτύχει. Στην κοινωνία μας, στην ήπειρό μας, είναι πολύ σημαντικό να είναι πρώτος, δεύτερος, τρίτος, δέκατο δεν έχει σημασία. Στην Ιαπωνία το πλαίσιο είναι διαφορετικό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να είναι κάποιος τελευταίος. Επομένω, τρώχουμε όλοι και δεν ενδιαφέρει να είναι κάποιο ε, πρώτο, αλλά να μην είναι τελευταίο. Και νομίζω ότι αυτό είναι το ευεδρικό σχέδιο. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ, κύριε Βίγια Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ε, στήριξή σας. Συμφωνούμε ότι η διαλειτουργικότητα είναι ο πλέον σημαντικός στόχος τον οποίο έχουμε θέσει. Αν κοιτάξουμε τις οικονομίες μας και κοιτάξουμε την απαιτούμενη ανάπτυξη και αν κοιτάξουμε την απαιτούμενη κινητικότητα για αυτή την ανάπτυξη, τότε συνειδητοποιούμε ότι δεν θα πρέπει να θεωρήσουμε τα, τους διάφορους τρόπους μεταφοράς ε, ως ανταγωνιστικούς αλλά ως συμπληρωματικούς. Η συμπληρωματικότητα λοιπόν παίζει καθοριστικό ρόλο. Αναφέρθηκα σε ένα από τα προγράμματα που μας απασχολούν. Έχουμε τον διάδρομο Ρότερνταμ, Τζένοβα, ε, τον σί ε, Αμβέρσα, Βασιλεία, λιον και Υπάρχει μια συμφωνία μεταξύ της ε, και του Βελγίου για σύνδεση Ρότερνταμ και ε, Αμβέρσα. Αυτό είναι η απαρχή του πλήρους ε, δικτύου που απαιτείται για τη μεταφορά εμπορευμάτων στην Ευρώπη. Έχω με αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα να απαντήσω σε ένα από τα ερωτήματα που έθεσε ε, η κυρία Γελασέντερ. Κάναμε ένα επιχειρηματικό σχέδιο για το διάδρομο Α. Απλά και μόνο για να παραθέσω ένα παράδειγμα. Αν συνδυάσουμε τα τρία μέτρα, πρώτον να εξετάσουμε και να βελτιστοποιήσουμε τις υποδομές, δηλαδή να κάνουμε όλες τις απαιτούμενες αλλαγές για τη βελτιστοποίηση των υποδομών. Δεύτερο, η εισαγωγή του RTMS και τρίτον, εναρμόνιση των κανόνων λειτουργίας. Για τη υπάρχουσα κατάσταση θα μπορούσαμε να έχουμε το στόχο να αυξήσουμε την ε, δυνατότητα κατά 50%, να μειώσουμε το κόστος κατά 20-30% και να αυξήσουμε την ασφάλεια κατά 20-30% επίσης. Συνεπώς αυτή είναι μεγάλη αριθμή, μεγάλα ποσοστά και με αυτή την άποψη πιστεύω ότι μολονότι ε, νιώθει κανείς απογοήτευση όταν είναι συντονιστής. Από την άλλη έχει πολλά κίνητρα γιατί μιλάμε για μεγάλους αριθμούς και για μεγάλη βαρύτητα του εγχειρήματό. Σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο ερώτημα του κυρίου Κράμερ για τα διαφορετικά συστήματα, είναι αλήθεια, υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος να βρεθούμε με 20 διαφορετικά συστήματα δεν, ε, αν ξεφύγει ο έλεγχος από τα χέρια μας. Η υπάρχουν συγκεκριμένες απαιτήσει για την ασφάλεια, ε, συγκεκριμένοι όροι στους διαγωνισμούς. Όλα αυτά θα πρέπει να εξαλειφθούν, να, επανα, να τα επαναδιαπραγματευτούμε με τις χώρες μέλη, έτσι ώστε να πάψει να υφίσταται αυτή η δυνατότητα. Από αυτή την άποψη φαντάζομαι ότι καταρχάς θα πρέπει να εναρμονίσουμε στο μέτρο του δυνατού τα πράγματα και να καλύψουμε τα κενά που υπάρχουν ή τον κίνδυνο δημιουργίας ε, κενών. Εάν δηλαδή τα κάνουμε αυτά, τότε θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε τον έλεγχο. Πώς θα το κάνουμε αυτό, θα το κάνουμε, όπως σας είπα, εναρμονίζοντας και τώρα βεβαίως συνειδητοποιούμε ότι το πιο σημαντικό πράγμα εδώ είναι οι δοκιμές. Χρειαζόμαστε μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική δοκιμών με εργαστήρια ε, που, επί των οποίων θα συμφωνήσουμε όλοι που είναι αποδεκτά σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αυτό είναι μία από τις βασικές προτεραιότητες κατά τη διάρκεια αυτής της εντολής να υπάρχουν κοινές ευρωπαϊκές διαδικασίες ελέγχου γιατί τότε μόνο θα είμαστε Είμαστε σίγουροι ότι θα υπάρξει προτυποποίηση παντού και δεν θα έχουμε προβλήματα όταν μετακινούμεθα από τη μία χώρα στην άλλη όταν διαχειρισχύσουμε την Ευρώπη. Έγινε ένα συγκεκριμένο σχόλιο ότι δεν αναφέρθηκα ποτέ στην, στον φορέα. Ζητώ συγγνώμη, συνεργαζόμαστε στενά με το φορέα έχουμε, αν σήμερα έχουμε ε, συγκεκριμένα πρότυπα, αυτό οφείλεται στο έργο της, ε, του ε, οργανισμού. Και αν τα καταφέρουμε και στο μέλλον, αυτό θα οφείλεται ε, στη συγκεκριμένο οργανισμό. Μην ανησυχείτε, συνεργαζόμαστε στενά και δίχως άλλο δεν μπορούμε να κάνουμε χωρίς τη δική τους βοήθεια. Ο κύριος Μπάγκερ έθεσε ένα ερώτημα για τα πρότυπα. Κατά πόσον οι χώρες έχουν τα ίδια πρότυπα. Κοιτάξτε, υπάρχουν διαφορές ιδιαίτερα για την ε, περίοδο ε, πριν. Πράγματι προτείναμε και γίνεται δεκτό από την Επιτροπή το να βοηθήσουμε και να υποστηρίξουμε τις χώρες που έχουν διαφορετικά πρότυπα. Να βοηθήσουμε να ε, φτάσουν στο πρότυπο 230D. Σε ό,τι αφορά την δημιουργία κινήτρων για την υιοθέτηση του συστήματος RTMS, κοιτάξτε, καταρχάς θα πρέπει να δείξουμε τι πλέον εκτίματα έχει και θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο σαφείς ε, στον τρόπο που επικοινωνούμε. Γνωρίζουμε ότι πράγματι η βασική περίοδος είναι η μεταβατική περίοδος της μετάβασης στην ε, πλήρη ε, εφαρμογή του ε, συστήματος διαχείρισης των χερσαίων, των δικών μεταφορών. Δεν είναι αρκετό όμως το να πείσει κανείς τους ε, σιδηροδρόμους. Έχουμε ένα πρόγραμμα, μάλλον επιδοτούμε και εάν είναι χαμηλό το τέλος ε, πρόσβαση στην περίπτωση του RTMS, νομίζω ότι αυτό θα καταφέρει να τους πείσει. Το σύστημα αυτό είναι υπό εξέταση στη Γερμανία. Νομίζω ότι δεν είναι αποτελεσματικό όμως. Είπαν, έχουμε δεσμευτεί στον διάδρομο A, να δούμε τι θα μπορούσαμε να κάνουμε. Σε ό,τι αφορά τους διαδρόμους δεν μπορούμε να δεσμευτούμε και συνεπώς αν ε, υπάρχει ο απαραίτητος εξοπλισμός, θα τους ε, χρηματοδοτήσουμε, θα τους επιδοτήσουμε για να τους δώσουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν το γερμανικό σύστημα στο γερμανικό δίκτυο. Τώρα, η γερμανική κυβέρνηση το να επιδοτήσει κάποιον για να καταστήσει γερμανικά συστήματα, γιατί δεν είναι έτοιμα να, να καταστήσουν το RTMS ε, ε, στο δικό του σύστημα. Κοιτάξτε, εγώ θα προτιμούσα τα χρήματα αυτά να τα πάρω και να τα επενδύσω ε, στο, σε ένα άλλο πρόγραμμα. Να λοιπόν που βρισκόμαστε. Νομίζω ότι έχουμε προχωρήσει, αλλά πολύ απέχουμε με τον τελικό στόχο. Όπως είπα, νομίζω ότι θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο και να γίνουν αποδεκτά όλα αυτά και να μπορέσουν να τεθούν σε εφαρμογή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ όλους θερμά. Δεν θέλω να ξαναρχίσω τη συζήτηση. Όχι, δεν απαντήθηκε η ερώτησή μου. Ήθελα τα πραγματικά νούμερα για την εγκατάσταση του RTMS στη Γερμανία, διότι είπατε ότι η Γερμανία κάνει λάθος. Ναι, ας μιλήσουμε για τα νούμερα και ας πάρουμε μία συγκεκριμένα περίπτωση, τον διάδρομο Α, για να ε, καταλάβετε το μέγεθος της απόφασης που θα πρέπει να ληφθεί για τα νούμερα. Καταρχήν στη Γερμανία μιλούσαμε για 4,5 δισεκατομμύρια. Αυτό αφορά όχι μόνο το RTMS, έχει να κάνει και με την ε, ανακαίνιση όλου του συστήματος interlocking. Ας πάρουμε τον διάδρομο Α Εφόσον το ATCS ε δεν έχει νόημα από μόνο του, θα πρέπει να ε, ανανεώσουμε ε, και τα, τις διασυνδέσεις interlocking. Για τι νούμερα μιλάμε λοιπόν. Εάν θέλουμε στο διάδρομο ένα, να ολοκληρώσουμε τις ε, συμπλέξεις, να εγκαταστήσουμε ε, το RTMS. Ε, αυτό σημαίνει 800 εκατομμύρια. Ένα πρόγραμμα που έχει νόημα από τεχνικής πλευράς είναι τα δύο τρίτα του διαδρόμου, να, στο, στα δύο τρίτα να ανανεωθούν οι συμπλέξεις και στο τελευταίο τρίτο να έχουμε ETCS. Αυτό σημαίνει 500 εκατομμύρια. Αλλά σήμερα στη χρηματοδότηση έχουμε διασφαλίσει μόνο 100 εκατομμύρια. Χρειαζόμαστε λοιπόν περαιτέρω 400 εκατομμύρια. Δηλαδή, για το διάστημα που προβλέπετε για <coughs> συγγνώμη, το διάδρομο Α, μιλάμε για 70 εκατομμύρια το χρόνο. Εάν κοιτάξουμε λοιπόν τα πλεονεκτήματα που προβλέπουν από το διάδρομο Α. Αν δούμε τι, το πώς έχουν δεσμευτεί η Γερμανία και οι άλλες χώρες που εμπλέκονται, ε, τα 77 εκατομμύρια είναι η δυσκολία που συναντάμε. Εκτός μικροφώνου είπε ο κύριος Κράμερ, κάτι δεν ακούσαμε. Ευχαριστώ κύριε Κράμερ, λέει ο πρόεδρος. Ευχαριστώ κύριε Βίνκ. Να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές για, την, ε, για τις πολύ πλήρεις εισηγήσεις τους και, τις, ε, και την ενδιαφέρουσα συζήτηση κατά την οποία απάντησαν ε, σε παρατηρήσεις και ερωτήσεις. Είμαστε ευγνώμονε, προσβλέπουμε στην καλή συνεργασία και στο μέλλον. Ελπίζουμε να σας ξαναδούμε. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Ευχαριστώ πολύ κύριε. Έτσι φτάνουμε στα διάφορα. Εάν ε, κάποιος βουλευτής έχει κάποιο θέμα για τα διάφορα θα τον πυροβολήσω, αλλά έπρεπε να ρωτήσω παρόλα αυτά. Δεν βλέπω να υπάρχει κανένα θέμα. Να σας θυμίσω ότι η επόμενη συνεδρίαση θα γίνει Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, λέει ο Πρόεδρος, στις 3. Ο Πρόεδρος ευχαριστεί ευγενικά τους διερμηνείς και εμείς ευχαριστούμε. Και ευχαριστώ φυσικά και τον Γιάννη, ο οποίος θα μας εγκαταλείψει τώρα. Πού θα χτυπήσω το σφυρί μου. Καλή τύχη λοιπόν.